Σας προτείνω να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, σας παρακαλώ. Σύμφωνα, μάλλον η ημερήσια διάταξη σας έχει διανεμηθεί, κανείς δεν πρόβαλε κάποια αντίρρηση για την ημερήσια διάταξη και τις ψηφοφορίες. Το μόνο συμπεριλαμβανικό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι θα πραγματοποιήσουμε μια συζήτηση κοινή για τα 5 και 6 Κρίστερσεν και Γιάρικ όπως το κάναμε και στην πρώτη άλλωστε ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε στο σημείο 2 που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 22 Φεβρουαρίου. Τα πρακτικά αυτά σας έχουν διανεμηθεί υπό την Προεδρία της κυρίας Λίντ. Μπορώ να πω τίποτα εγώ για αυτά τα πρακτικά, αλλά εντάξει, αλλά επειδή δεν άκουσα να προβάλλετε και κάποια αντίρρηση, σας προτείνω να εγκριθούν τα πρακτικά αυτά. Πάμε παρακάτω, οι ανακοινώσει της Προέδρου, σημείων 3. Όσα θα ήθελα να σας πω, αλλά είναι τρία αυτά. Πρώτα απ' όλα, στους φακέλους σας θα δείτε τα πράγματα σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων με την Ισπανική Προεδρία στις 27 Ιανουαρίου. Την έχετε σε τρεις γλώσσες ε, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, την ανακοίνωση αυτή. Και επίση ε, θα δείτε κάτι παρόμοιο, την ανακοίνωση, δηλαδή για την αντιπροσωπεία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και αυτό στα πλαίσια των εργασιών των Εθνών 3-7 ε, Φεβρουαρίου του 2010 η ιδέα ανακοίνωση αυτή είναι διαθέσιμη σε τέσσερις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά τελευταία μου ανακοίνωση για τα πρακτικά του άτυπου συμβουλίου ΕΠΣΚΟ στη Βαρκελόνη 28-29 Ιανουαρίου. Συμμετείχα δε και εγώ εκπροσωπώντας εδώ την Επιτροπή σε ένα μέρος των εργασιών και τουλάχιστον ε, το έχετε αυτό στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά και στα ισπανικά. Αν δεν υπάρχει τώρα από εσά κάποιο άλλο σημείο που θέλετε να θίξετε για τις εργασίες μας, να πάμε στο σημείο 4. Ποιο είναι το σημείο 4? Οι τροπολογίες ε, από ε, την κυρία Ρεζίνα Μπεστός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνεχή για τις γενικές διατάξεις, για την απλοποίηση διαφόρων απαιτήσεων και διατάξεων για την δημοσιονομική διαχείριση. Είχαμε ζητήσει την ενισχυμένη συνεργασία σε αυτό το θέμα και δυστυχώς ε, μια απλή διαδικασία γνωμοδότησης αυτή να έχουμε και η επί της ουσίας είναι η Περιφερειακών Υποθέσεων Επιτροπή και υιοθέτησε τη γνωμοδότηση στην συνεδρίασή της στις 17 και 18, μάλλον θα το κάνει 17-18 Μαρτίου. Είχαμε 27 τροπολογίες για την έκθεση της κ. Μπάστος και έχετε εσείς το λόγο για να δούμε τι γίνεται με, αυτά, με αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες και οι οποίοι με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη βελτίωση της γνωμοδότησης την οποία εγώ εκπώνησα. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας θα βοηθήσει να υπάρξει μεγαλύτερη απλοποίηση της πολιτικής συνοχής, να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η πολιτική με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και επομένως να βοηθήσει τη διατήρηση και τη δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας στα κράτη-μέλη. Για τις τροπολογίες λοιπόν αυτές, συμφωνώ με τις τροπολογίες 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21 και 26. Οι 5 έχει σαν στόχο καλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 2020 υπέρ του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής τροπολογία 7 υποστηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι βιώσιμες η 8 έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η 9 αφορά την παρουσίαση από την Επιτροπή στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μιας έκθεσης διακόπτεται η ομιλήτρια. Ίσως πιο αργά αν θέλετε λέει η Πρόεδρος γιατί αλλιώς δεν θα σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Νομίζω, νόμιζα ότι ακολουθούσα ένα εφικτό ρυθμό ομιλίας. Η τροπολογία 10 λοιπόν συνάπτεται με τις επιχειρήσεις και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης από τις επιχειρήσεις. Η 11 υπογραμμίζει τη σημασία του να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα επιτρέψουν στο κοινωνικό ταμείο να έχει ταχεία αντίδραση σε εποχές κρίσης για να αποφύγει καθυστέρηση στην εκτέλεση των προγραμμάτων. Η τροπολογία 12 έχει να κάνει με την βέλτιστη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια καλύτερη εφαρμογή των ε, ενεργών μέτρων στην αγορά εργασίας. Η 13 έχει να κάνει με την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων, χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η 14 προβλέπει μια παράταση της προθεσμίας για την ε, αυτόματη ακύρωση των ε, ε, πιστώσεων που έχουν ξεκινήσει από το 2007 λόγω της ε, καθυστερημένης έγκρισης των προγραμμάτων. Η τροπολογία 16 έχει να κάνει με το περιβάλλον και μάλλον το πλαίσιο εργασίας των ατόμων με αναπηρίες. Η 21 έχει να κάνει με αυτά τα οποία είπαμε με τον εισηγητή της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων και έχουν γίνει δεκτές από το Συμβουλίο. Όλες αυτές οι τροπολογίες λοιπόν και 26 μαζί με 21 συμβάλλουν στην έκθεση αυτή, γι' αυτό τις υποστηρίζουμε. Είμαι εναντίον τώρα στις τροπολογίες 6, 15, 17, 19 και 20. Στην 6 γιατί μειώνει τη σφαίρα εφαρμογής των πόρων αυτών των χρηματοοικονομικών που έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχή. Είμαι εναντίον στις 15 γιατί τα, οι μικροπιστώσεις δεν πρέπει να επισέρχονται μέσα στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, εναντίον της 17, γιατί αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού με έναν τρόπο που δεν πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος, κατά της 18, γιατί δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία τα στατιστικά, και η 19 και 20 γιατί δημιουργούν προβλήματα σε ήδη χρηματοδοτούμενες ενέργειες οι οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν άρδιν. Επομένως, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτές τις σύντομες και συνοπτικές ελπίζω παρατηρήσεις. Νομίζω ότι σας έχω δώσει μια πλήρη εικόνα σε σχέση με τα διακυβευόμενα σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και τους στόχους της γνωμοδότησης που εγώ έχω εκπονήσει, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τις συστάσεις και τις προτάσεις των συναδέλφων μέσω των τροπολογιών και πάλι θέλω να, συ... να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συμβολή τους. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Μήπως κάποιος άλλος θα επιθυμούσε το λόγο τώρα. Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος ε, ενός συναδέλφου ο οποίος είναι σε ταξίδια αυτή τη στιγμή, κύριε Τσίπε, θα ήθελα να δώσω τη δική του άποψη για τα θέματα αυτά. Τη στιγμή που έχουμε την ε, οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, η προκαταβολική χρηματοδότηση κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολύ καλή ιδέα, δυστυχώς. Το Συμβούλιο έχει ήδη πάρει απόφαση πριν ακούσει την άποψη του Κοινοβουλίου και έχει πάρει μια θέση διαφορετική από αυτή την οποία υποστηρίζει η Περιφερειακή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένω, αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα εμεί να επιμείνουμε σε μια χρηματοδότηση, προχρηματοδότηση κατά 100%. Γιατί δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει μια τέτοια απόφαση. Έχει περάσει πολλής χρόνος ήδη και επομένως εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία με την μεταφορά ε, κονδυλίων που δεν έχουν ήδη μεταφερθεί βάσει του άρθρου 207. Αυτή είναι λοιπόν η, η παρατήρηση που θέλω να κάνει ο συνάδελφός μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Φιγερέντο. Εγώ δεν έχω καταθέσει αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση τροπολογίας, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτήν την ιδέα του, της χρηματοδότησης κατά 100% για τις χώρες οι οποίες έχουν υψηλό επίπεδο ανεργίας. Το να μην υπάρχει απέτηση συγχρηματοδότησης για αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας, σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Αυτό για μένα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο στην τρέχουσα φάση της κρίσης. Ξέρω ότι όλα αυτά σημαίνουν και απώλεια χρόνου. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού, των κανονισμών αυτών, αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι απαραίτητο από τη δική μας πλευρά να εξακολουθούμε να ασκούμε πίεση προς το Συμβούλιο για να λειτουργήσει ο στόχος αυτός της χρηματοδότησης κατά 100%. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς οι οποίοι θα διευκολύνουν την κατανομή των πόρων και την σωστή χρησιμοποίησή τους και επίσης την ε, καλύτερη εκμετάλλευση των πλεονασμάτων από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θέλω να επιμείνω στο ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση της ανάγκης συγχρηματοδότησης για μια χρονική περίοδο όπως αυτή της κρίσης, ιδίως για τις χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Γιατί αλλιώς, αντί τα ταμεία αυτά να βοηθούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή, υπάρχει ο κίνδυνος τα ταμεία αυτά να επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο τις ανισότητες και τις αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών για τα κάτι μέλη τα οποία δεν θα έχουν τη δυνατότητα συγχρηματοδότηση, απλώς και μόνο δεν θα χρησιμοποιούν τα ταμεία αυτά, ενώ οι άλλες χώρες οι οποίες θα έχουν χρήματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα ταμεία. Αυτό τελικά θα οξύνει ακόμα περισσότερο τις εδαφικές, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και δεν θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή που είναι ο κύριος στόχος αυτών των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θα επιθυμούσε τώρα να λάβει το λόγο. Η εισηγητριά μας και πάρα κύριε Μπαστός έχει το λόγο. Μέχρι τώρα μπόρεσε ήδη να δει τι γίνεται για τη συνεργασία με την Επιτροπή που είναι ορμόδια από τις γιατί θα κάτι τέτοιο θα ήταν τρομερά σημαντικό και για να μην ε, και να ξεσπάσουμε και το μέλλον ακριβώς, να δούμε στο θέμα αυτό όχι μόνο συμβολικά, αλλά θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια συνεργασία πραγματική και να λάβουν υπόψη τις τροπολογίες ε, στην Νομική Επιτροπή. Τώρα, αν έχετε κάτι να μας πείτε και να σας ενημερώσετε, θα σας ευχαριστούσαμε. Θα θέλαμε να τα ακούσουμε αυτά. Πέρα από αυτό όμως εγώ σας προσκαλώ και θα σας κινητοποιήσω όσο γίνεται η Νομική Επιτροπή να αποδώσει μια κάποια σημασία στη δική μας τη βοήθεια πάνω στο θέμα αυτό. Γνωρίζετε όλοι σας ότι πίσω από αυτά υπάρχει μια επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε γι' αυτό και η συνδιάσκεψη των Προεδρών ε, πήρε μια απόφαση, δεν συμφωνώ, αλλά μας επιβάλλεται αυτή, με αυτή θα πρέπει να συμβαδίσουμε, τουλάχιστον να βελτιώσουμε να γίνεται περισσότερο τη δυνατότητα παρέμβασής μας σε αυτά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια μας την κυρία Μπαστός, μήπως κάποιος άλλος θα επιθυμούσε τον λόγο, όχι η εισηγήτρια λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους οι οποίοι παρενέβησαν για τις τροπολογίες και εξήγησαν ποια ήταν η άποψή τους και ο στόχος των τροπολογιών που έχουν καταθέσει ή σε μια συγκεκριμένη περίπτωση για την μη παρουσίαση τροπολογιών σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, χρηματοδότησης κατά 100%. Νομίζω ότι το συμπέρασμα ήταν για πολλούς ότι η χρονική στιγμή παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να χρονοτριβήσουμε και να χάσουμε χρόνο για να επιτύχουμε το στόχο αυτό του 100% συγχρηματοδότησης, μάλλον χωρίς χρηματοδότηση, 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το ουσιαστικό είναι να μπορέσουμε να επιτύχουμε το ταχύτερο δυνατόν του οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους αντιμετώπιση της κρίσης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Σε ό,τι αφορά <clears throat> τη βασική φιλοσοφία που αφορά την τη συγχρηματοδότηση ή τη χρηματοδότηση κατά 100% αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον και έθεσε και η πρόεδρός μας το ερώτημα του κατά πόσο αν εγώ είχα διαπραγματευτεί με την ε, Επιτησίλη αρμόδια επιτροπή, την Περιφερειακή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το, τη μεταρρύθμιση της φιλοσοφίας των, κοινοτικών των ταμείων, του, του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. Εγώ ακόμα δεν έχω προβεί σε αυτές τις ενέργειες, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει. Εμείς σαν Επιτροπή Απασχόλησης επομιζόμαστε μια μεγάλη ευθύνη, μια συνυπευθυνότητα στον τομέα αυτό. Εγώ είμαι φυσικά απόλυτα διαθέσιμη να προχωρήσω σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις με την αρμόδια Επιτροπή επί της ουσίας, δηλαδή Περιφερειακή. Και θα ήθελα εδώ επίσης να πω ότι αυτό το οποίο αποφασίστηκε από το Συμβούλιο διαπνέεται από ένα πραγματιστικό πνεύμα, δηλαδή να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τους οικονομικούς πόρους που είναι στη διάθεσή τους το ταχύτερο δυνατό. Εγώ κατανοώ λοιπόν και υποστηρίζω την πραγματιστική αυτή στάση που είχε η σοσιαλιστική ομάδα για το θέμα αυτό και που δεν κατέθεσαν καθόλου τροπολογίες οι οποίες ζητούσαν να, διαπραγματευθούν, να συνεχίσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σε σχέση με την επίτευξη του στόχου της χρηματοδότησης 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Κατανοώ ότι έχετε διάθεση να συνεργαστείτε με την Περιφερειακή Επιτροπή. Δεν πρέπει να είναι όμως κανείς διαθέσιμος. Θα πρέπει να τον διακρίνει και κάποια έτσι, ας το πούμε, επιθετικότητα για να κερδίσει και κάτι βέβαια διπλωματικά και ευγενικά να γίνει αυτό. Γιατί η Περιφερειακή Μισοτροφή δεν μας ακούει και τόσο γι' αυτό θα πρέπει κάπως να την πιέσουμε. Για το τελευταίο σημείο που θίξατε εσείς, Όλοι ήταν ήσυχοι και ήρεμοι και κανεί δεν ξανά άνοιξε το θέμα αυτό για αυτή τη χρηματοδότηση 100%. Αυτό έχει να κάνει ακριβώ με τι εξηγήσει που έλαβαν όλοι από τότε και η σχετική διευκόλυνση ήταν προσωρινή φύσεως μόνο και σε σχέση με τον προπολισμό των κρατών μελών. Ο κύριος στόχος που ήταν να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη σε παρόμοιες φάσεις κρίσης. λοιπόν παίρναμε φόρα για να επιδείξουμε μακρύτερα και αυτό σχετικά με την πλήρη ανάληψη της χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγείται κάπως ε, έτσι και το ισχνό ενδιαφέρον το αρχικό τουλάχιστον της Επιτροπής. Είναι από τα σημεία πάντως που θα πρέπει να τα δούμε, να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε, να τα σωματώσουμε. Δεν θα αποτελέσει βέβαια την κατευθυντήρια γραμμή αυτής της πολιτικής, αλλά και χρειάζεται να το προσέξουμε. Θα πάμε για τα ελληνικά πράγματα στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μελλοντικά σε μια παρόμοια περίπτωση δεν θα χρηματοδοθεί 100% ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Χρειάζεται να αλλάξουν οι προπολογισμοί, ο προϋπολογισμός ε, βέβαια βαριέ μετασχηματισμό αυτό, αλλά ο τρόπο με τον οποίο συζητήσαμε τότε σχετικά με την έκθεσή σα για το θέμα αυτό θα μπορούσε να μα οδηγήσει να ξαναξεκινήσουμε αυτό το διάλογο και να κρατήσουμε αυτά τα θέματα, να τα συλλογιστούμε καλύτερα για τι μελλοντικέ μα εργασίε. Ευχαριστούμε λοιπόν την εισηγήτρια θα ψηφίσουμε για τις τροπολογίες αυτές αρχικές τις οποίες καταθέσατε εσείς και μετά τις υπόλοιπες που κατατέθηκαν τους συναδέλφους ε, στη συνάντησή μας. Αύριο θα γίνει αυτό. Τελειώσαμε το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Ε, πάμε παρακάτω. Πάμε στο σημείο 5. Και το λόγο έχει ο κύριος Όλε Κρίστενσεν. Ε, έφτασε, ήλθε το θέμα είναι 68 τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, από την Οικονομική Κοινωνική Τυπή για τις για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει, για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τις πράξεις επανατιτλοποίησης και τον υποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών. Ε, έχει το λόγο εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία, η οποία ήταν θαυμάσια. Θα είμαι πολύ σύντομος. Έχουμε καταθέσει συμβαστικές τροπολογίες, αλλά δεν συμφωνούμε με όλες τις τροπολογίες. Υπάρχουν δύο ειδικά δέσμες τροπολογιών ή μάλλον δύο τομείς επί των οποίων δεν μας αρέσουν οι τροπολογίες το μεταβλητό τμήμα καταρχάς των πόνους. Επανεξέτασα το κείμενο για να δω ότι όλα συνάδουν με αυτά που αποφασίσαμε στη συνεδρίασή μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μιλάμε και για μια επιτροπή που θα πρέπει να υπάρχει στις μεγάλες τράπεζες. Γίνεται λόγος και για αυτό το θέμα. Αυτό νομίζω ανταποκρίνεται σε αυτό που αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Πίτσμπουργκ. Τώρα, τα μπόνους. Για το μεταβλητό τμήμα των μπόνους. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Δεν θέλουμε το μεταβλητό των πόνους. Αλλά στη Σύνοδο Κορυφής ε, του Πίτσμπουργκ επίσης αποφασίστηκε κάτι τέτοιο. Συμφώνησε το Συμβούλιο. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να ξαναδούμε αυτά τα δύο σημεία. Υπάρχουν έπειτα και κάποιες μικρές λεπτομέρειες που θα ήθελα να αναφέρω. με τους διάφορους συντάκτες θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα για να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από την αυριανή ψηφοφορία. Έπειτα, πρέπει να συζητήσουμε και για τα πράγματα επί των οποίων συμφωνούμε. Είναι τα περισσότερα αυτά. Είμαι πεπισμένος ότι θα συνεισφέρουμε πολύ επικοδομητικά στην γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής. Και ελπίζω η Οικονομική Επιτροπή να λάβει υπόψη της την, το κείμενό μας, την έκθεσή της. Ευχαριστώ επίσης τη Γραμματεία, με την οποία είχα μια θαυμάσια συνεργασία, με βοήθησε πάρα πολύ και θα ακούσω με μεγάλη προσοχή τα όποια σχόλιά σας. Κανένας από την ε, Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο για αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν πρέπει... να δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Λεϊάρικα. Δεν θέλω να ανακατέψουμε τις διαδικασίες. Θέλω τώρα να συζητήσουμε τους συμβιβασμούς και τις τροπολογίες. Πάτρικ, συγγνώμη. Αντίθετα από ό,τι είχα πει στην αρχή, καλύτερα να διεκπαιρεώσουμε την έκθεση Κρίστενσεν και μετά τη δική σας έκθεση. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε να μιλήσετε, αν θέλετε να μιλήσετε για την έκθεση Κρίστενσεν, κύριε Λεγιαρίκα, μπορείτε καλύτερα να πάρετε το λόγο. Ο Τόμας Μαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πάρω θέση για την έκθεση Κρίστεν. Είχαμε την ευκαιρία στην τελευταία εβδομάδα, προηγούμενη εβδομάδα του Στρασβούργου να συζητήσουμε για τα θέματα των συμβαστικών τροπολογιών και βρήκαμε πολλά σημεία στα οποία μπορεί να υπάρχει γενική υποστήριξη και άλλα σημεία με τα οποία μπορούμε να ζήσουμε. Τώρα, σε ορισμένα σημεία δεν έχουμε βρει κάποια λύση. Εξακολουθούμε να είμαστε εναντίον των ανεξαρτήτων επιτροπών για τις αμοιβέ. Εξακολουθούμε επίσης να έχουμε προβλήματα με την τροπολογία υπαριθμών 2, η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει μονάχα τις τροπολογίες των αριστερών ε, και του αριστερού κόμματος και όχι τις δικές μας τροπολογίες. Επίσης, στην τροπολογία υπαριθμών 10, υποστηρίζουμε την ε, μεταβλητότητα των αμοιβών. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό της στρατηγικής αμοιβών των επιχειρήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης το σημείο Δέλτα, όπου υπάρχει μια αλλαγή στον ορισμό των ε, managers, μπορούμε να το δεχτούμε και στο σημείο ε έχουμε προτείνει να υπάρξει μια θετική υποστήριξη γιατί αυτό υποστηρίζει τα Ευρωπαϊκά Εργασιακά Συμβούλια. Για άλλες τροπολογίες τώρα έχω την υποστήριξη από το κόμμα μου για άλλες όμως δεν έχω αυτή την υποστήριξη Είμαστε εναντίον της Α και της Β των συμβαστικών αυτών τροπολογιών αυτή είναι η θέση του ΕΛΚ αλλά για την Σ, Δ και Ε έχουμε πλήρη υποστήριξη Νομίζω ήταν πολύ καλή η συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κρίστενσεν Υπήρχαν ορισμένες θέσεις, οι οποίες εμείς δεν μπορούσαμε να αποδεχτούμε, παρά τις αλλαγές. Λοιπόν και παρά το γεγονό ότι ορισμένε τροπολογίε δεν τι δεχόμαστε, νομίζω ότι είναι μια έκθεση η οποία είναι ισορροπημένη και ίσω πρέπει να τη συνδυάσουμε και με την επόμενη έκθεση, γιατί και για τι δύο εκθέσει θα πρέπει να ξεβρεθεί μια κάποια ισορροπία. Αυτή είναι η θέση και τη δική μου ομάδα. Θα ήθελα κάποια πράγματα να αλλάξουμε, βέβαια, αλλά ακόμα και χωρί να αλλάξουν νομίζω ότι μπορεί να είναι αποδεκτή η κατάσταση μερικές φορέ η ελπίδα είναι πιο δυνατή από τι αρχέ και την πραγματικότητα. Euh, euh, Κύριε την όταν λέτε να μετακινηθούμε, τι σημαίνει αυτό. τάσει ε, τροπολογιών. Δεν θέλετε τι τροπολογίε. Είσαστε μεταξύ των δύο. Πού ακριβώ είστε. Το να κινηθούμε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλε τα καταφέρνει πολύ καλά. Κάνει συμβιβαστικέ προτάσει, είτε μπορούμε να τι δεχτούμε ή όχι. Τώρα, αν το ΕΛΚ μπορεί να δεχτεί τι τροπολογίε C, D και Ε, θα μπορούσε, αν είχε κινηθεί περισσότερο εισηγητή, να δεχτεί και την Α και την Β. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούσε να το κάνει. Την C, την Τζ και, τε, και την Ε, e, τι έχουμε δεχτεί όπω και τι περισσότερε τροπολογίε. Την Α και την Β όμω δεν μπορούμε να τι δεχτούμε ε, πρέπει να καταλάβουμε τι εννοείται τώρα με αυτά που λέτε, έτσι, δεν καταλάβουμε ακριβώ ε, ποιο είναι το διακύβευμα εδώ, τι παίζεται εδώ. Φαντάζομαι όμως ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές το πιασαν το νόημα. Η κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ τον κύριο Κρίστενσεν για τη δουλειά του που τον ευχαριστώ που ενέπλεξε όλες τις πολιτικές ομάδες και κυρίως τους πράσινους για τις συμβαστικές τροπολογίες που δεν ήταν καθόλου εύκολες να υλοποιηθούν. Θα τονίσω ότι λυπόμαστε που δεν πήγαμε αρκετά μακριά, ιδίως ε, στο θέμα των ε, μπόνους ε, την προθεσμία από τρία σε πέντε χρόνια ε, μέσα στην οποία θα μπορούσε να αναβληθεί η πληρωμή, η καταβολή τους. Αλλά έχουμε σημαντικά σημεία πρόοδου για τις τροπολογίες ε, της πράσινης, την απαγόρευση των μεταβλητών αποδοχών, ε, την, την εμπλοκή των εργαζομένων στην εκπόνηση των πολιτικών για τις αποδοχές, την δημιουργία επιτροπών ε, απολαβών για ανεξάρτητες μάλλον και ασχολούνται επίσης αυτές οι επιτροπές ασχολούνται με τις ε, κοινωνικές και περιφερειακές ευθύνες των εταιριών. Νομίζω ότι αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες νομίζω θα περάσουν πλειοψηφία και θα μπορούσαμε να πιέσουμε την Οικονομική Επιτροπή, ούτω ώστε οι δικέ μα προτάσει να μην μείνουν γράμμα κενό περιεχομένου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για την συμβαστική τροπολογία Α. Ο Τόμας Μάν μίλησε για την διάθεση μετακίνησης. Ε, ίσως υπάρχει μια δυσκολία ε, για το θέμα των αποδοχών. Στην προηγούμενη ζωή μου έμαθα ότι αυτές οι επιτροπές για τις αποδοχές ήταν κάτι το οποίο συζητιόταν. Ήταν μεταξύ των θεμάτων της πρώτης έκθεσης που μιλούσε για θέματα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ πριν την εποχή Μπαρόζο. Μιλάμε για την έκθεση Winter, όπου η εφαρμογή και η δημιουργία τέτοιων επιτροπών ε, είχε ήδη προταθεί στην έκθεση αυτή. Μετά, ε, στην προσπάθεια να δώσουμε απαντήσεις στην κρίση ε, και στα πλαίσια της Βασιλείας, συζητήσαμε το θέμα της διάρθρωσης εποπτείας των κινδύνων και αξιολόγησης των αποδοχών. Και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Για να μην υπάρχουν υπερβολικές... Ε, να μην προβαίνουν τα στελέχη των επιχειρήσεων σε προχωρούν σε υπερβολικά ρίσκα, ας πούμε. Επίσης, όπως είπε και ο εισηγητής στο Pittsburgh, είπαμε κάποια πράγματα. Βέβαια, οι Αμερικανοί υπαναχώρησαν σε σχέση με τι δεσμεύσει Πίτσμπουργκ. Γιατί λοιπόν εμεί να μην το κάνουμε επίση. Αλλά στο Pittsburgh εμεί ήμασταν αυτοί που θέσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτά τα στοιχεία. Θα ήταν λοιπόν παράδοξο εμεί οι ίδιοι να μην σεβαστούμε τι δεσμεύσει που ζητήσαμε να αναλάβουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό το θέμα της Επιτροπής για τις αποδοχές υπάρχει σαφώς στα συμπεράσματα του G20 του Pittsburgh που είναι ένα μικρό βήμα για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των επιχειρήσεων. Τώρα δεν ξέρω πώς, τι, τι, ισορροπίες δημιουργούνται, αλλά θα ήθελα να ξαναδούμε το θέμα αυτό. Το θέμα της τροπολογίας, της συμβαστικής τροπολογίας Α. Πολλό δε μάλλον που αυτό το θέμα στις συζητήσεις με τους εργοδότες δεν είναι και τόσο ταμπού. Ορισμένοι εργοδότες, ορισμένα συνδικάτα εργοδοτών συνειδητοποιούν ότι πρέπει να δεχτούν αυτή την πρόταση. Η πάση δεν είναι απρόθυμη. Υπάρχουν δηλαδή σημεία πρόοδου σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήταν λοιπόν κρίμα για την έκθεση Κρίστενσεν να μην περάσει αυτή η τροπολογία. Αυτή η συμβιβαστική τροπολογία. Ε, άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο. Αν όχι, θα δώσω το λόγο ξανά στον εισηγητή για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ, λέει ο εισηγητής για τις παρατηρήσεις σας. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και στις δύο τελευταίες αυτές την Α και την Β συμβαστικές τροπολογίες. Δεν ξέρω, ίσως με τον Τόμας Μαν θα μπορέσουμε να συναντηθούμε και πάλι σήμερα το απόγευμα και ενδεχομένως να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τις δύο αυτές επίμαχες τροπολογίες. Εγώ θέλω να προσπαθήσω αν είναι δυνατόν. Τρέμπιεν λέει η πρόεδρος, αν βγείτε και οι δύο από την αίθουσα, τότε στο τέλος δεν θα υπάρξει και πολλοί κόσμος για να παρακολουθήσει συνέχεια των εργασιών μας. Θα ψηφίσουμε αύριο για το σχέδιο αυτογνωμοδότησης. Και σας προτείνω ως εκ τούτου να προχωρήσουμε στην έκθεση του κυρίου Λεϊαρίκ, επί του οποίου κειμένου υπάρχουν και πάλι πέντε συμβαστικές τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω στον εισηγητή τις εργασίες της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, γιατί εμείς γνωμοδοτούμε έναντι της νομικής επιτροπής. Και η έκθεση του κυρίου λένε, δυστυχώς είναι μονάχα, λένε στα αγγλικά διαθέσιμη. Και έχει κατατεθεί πολύ καθυστερημένα αυτή η έκθεση. Στις 4 Μαρτίου μονάχα κατατέθηκε. Και θυμάστε ότι όταν εξετάσαμε για πρώτη φορά την έκθεσή σας, ένα από τα πράγματα τα οποία μας απασχολούσαν είναι να εξασφαλίσουμε ότι η σφαίρα εφαρμογής της έκθεσης πρωτοβουλίας του κυρίου λένε είναι, να είναι ακριβώς αυτή η σφαίρα εφαρμογής που μας ενδιαφέρει εμάς ως Επιτροπή Απασχόλησης. Δεν ξέρω λοιπόν αν εσείς από τη δική σας πλευρά είχατε τη δυνατότητα να εξετάσετε το κείμενο βάσης σε σχέση με το οποίο εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε και να το συμπληρώσουμε και να το βελτιώσουμε. Αλλά μέχρι αύριο νομίζω θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώ τι λέει το αρχικό κείμενο, προτού ψηφίσουμε καν τη δική σα γνωμοδότηση. Κύριε και έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε τι συμβαστικέ τροπολογίε, ακόμη και τι τροπολογίε που ενδεχομένω να μην καλύπτονται από τι συμβαστικέ τροπολογίε. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετέσχουν στη σύνταξη αυτής της νομοδότησης και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι καταλήξαμε σε μια καλή συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι, ΕΛΚ, Πράσινοι, ε, Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Για τις τροπολογίες θα τις χωρίσω σε επιμέρους θέματα. Οι τροπολογίες 4, 5 και 6 αφορούν την ευθύνη του τωρινού συστήματος και μοντέλου ε, αμοιβή σε ό,τι αφορά την ανάληψη κινδύνων. Όλα αυτά τα έχουμε συνδυάσει στη συμβαστική τροπολογία Α που τονίζει ότι τα κέρδη τα οποία προβλεπόταν είχαν να κάνουν με τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία χωρίς να λάβουν υπόψη την πραγματική οικονομία και τα προβλήματα απασχόληση. Γι' αυτό το λόγο εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω τις τροπολογίες 8 καθώς και 9 γιατί ο αντίκτυπος αυτού του συστήματος αμοιβή στην πραγματική οικονομία υπήρξε αρνητικός. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 11, 12 καθώς και 13 βρίσκονται στα πλαίσια συμβεστική τροπολογίας Β ζητούν να υπάρξει μια νέα χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική, η οποία να βασίζεται σε εποπτικούς και δεοντολογικούς κανόνες και να υπόκειται σε εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές που να έχουν δεσμευτική εξουσία. Τονίζεται ότι η Επιτροπή μας απασχόληση με τον τρόπο αυτό δίνει ένα σαφές μήνυμα υπέρ της δημιουργίας μιας εξουσίας που θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και θα εξασφαλίζει τη ρύθμιση στο χρηματοοικονομικό τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάται και σε άλλου χώρου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου εξάλλου. Γι' αυτό το λόγο εγώ υποστηρίζω τι τροπολογίε 27 καθώ και 28 τη κυρία Περέ, η οποία υποστηρίζει μια τέτοια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα. Τροπολογίε 14 και 15 υπενθυμίζουν ότι η Κομισιόν είχε κάνει στις 30 Απριλίου του 2009 ήδη κάποιες συστάσεις, όλα αυτά περιλαμβάνουν συμβαστική τροπολογία σε λατινικό, Εκεί τονίζουμε ότι υπάρχει και μια ευθύνη των επιχειρήσεων έναντι του κοινωνικού περίγυρου και του περιβάλλοντος, αυτά στις τροπολογίες 16 και 17 του κύριου Κοφεράτη και επίσης στις τροπολογίες 25 και 26 που έχουν συγχωνευτεί στη συμβαστική τροπολογία ε. Η κοινωνική ευθύνη συνδέεται επίσης με τον αγώνα κατά όλων των διακρίσεων, όπως τονίζει η τροπολογία 32, μέσα στα οποία περιλαμβάνεται η ισότητα αποδοχών ανδρών και γυναικών, που είναι η τροπολογία 34 και υποστηρίζω λοιπόν αυτή την τροπολογία. Υπάρχει το θέμα της αμοιβή που αφορά τροπολογίες από το 18 το 24. Προτείνω να τις συνενώσουμε αυτές στην συμβαστική τροπολογία ΔΕΛΤΑ, ΔΕ λατινικό. Και εξάλλου πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι για να τονίσουμε ότι οι αμοιβέ των ανώτερων στελεχών είχαν αρνητικό αποτέλεσμα γιατί οδήγησαν σε αλόγιστη ανάληψη κινδύνων ότι πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν αυτές οι αμοιβέ διαφόρων ειδών και όχι μονάχα οι μισθολογικές αποδοχές αλλά και τα άλλα πριμ και μπόνους, τα λεγόμενα χρυσά αλεξίπτωτα, οι προαιρέσεις για αγορά μετοχών κτλ. Και ιδίω αυτό σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τύχει αρρωγής από τα κράτη-μέλη ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίση αυτά τα εισοδήματα των στελεχών να φορολογηθούν με τον τρόπο που προβλέπεται στα κράτη-μέλη για να μην υπάρξει ένα σύστημα δύο μέτρων και δύο σταθμών σε ό,τι αφορά το εισόδημα, την πρόσοδο από την εργασία και την πρόσοδο από την χρήση κεφαλαίου. Όπως λέει επίσης η τροπολογία 36 του κ. Μπαλταζέρ και της κυρίας Μεσνέρ από το ΕΛΚ, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της εργασίας προς όφελος της ε, πραγματικής οικονομίας που έχουν ένα θεμελιώδη χαρακτήρα, το προσυπογράφει και εγώ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα έσοδα από αυτήν την φορολόγηση των αποδοχών των στελεχών θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την υποστήριξη της απασχόλησης και των δημοσίων υπηρεσιών που δοκιμάζονται από την χρηματοοικονομική κρίση αλλά που πρέπει συγχρόνως να θεωρηθούν ως εργαλεία κατά της κρίσης κατά την άποψή μου το θέμα των αποδοχών και συγχρόνως το θέμα της ευθύνης έναντι του περιβάλλοντος και του κοινωνικού χώρου είναι θέματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στα τεκθενόμενα. Γι' αυτό δεν υποστηρίζω τις τροπολογίες 41-42 που λένε ότι απλώς θα πρέπει να παραμείνουμε στο τωρινό πλαίσιο διαβούλευσης και συμμετοχής. Αντίθετα πιστεύω ότι τα συνδικάτα χρειάζονται περαιτέρω δικαιώματα τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν μια αυξημένη, ένα αυξημένο ανταγωνισμό. Γι' αυτό υποστηρίζω τις τροπολογίες 39 και 40 που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και που συνδέουν την ε, αμοιβή των στελεχών με επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν και θα διατηρήσουν θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε επίπεδο επιχειρήσεων, γι' αυτό έχω καταθέσει τροπολογία 25, η οποία δημιουργεί ένα πολυετές πλαίσιο τουλάχιστον τριών ετών, προτού εκτιμηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος των αποφάσεων οι οποίες θα έχουν ληφθεί και θα μπορούσε να υπάρχει αντίκτυπος στις αποδοχές, αν είναι αρνητικός και ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών. Γι' αυτό υποστηρίζω την τροπολογία 46 του κ. Σομπόρ σε σχέση με το, την θέση ανώτατου ορίου και την ενδεχόμενη απαγόρευση περαιτέρω πριν κτλ. Λυπάμαι τώρα που η διαπραγμάτευση των συμβαστικών τροπολογιών έγινε σε βάρος της ιδέας μιας ιδέας πιο προοδευτικής για το μεταβλητό τμήμα των αποδοχών. Πρέπει να υπάρξει ισότης σε ό,τι αφορά την φορολόγηση των προσόδων της εργασίας και των προσόδων του κεφαλαίου. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και καταδεικνύει η κρίση ότι η φορολόγηση του κεφαλαίου σε υψηλότερο επίπεδο από ότι η φορολόγηση των προσόδων της εργασίας είναι απαραίτητη για την κοινωνική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αλλά και για την κοινωνική και για την οικονομική αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας λοιπόν. Ευχαριστούμε. Κυρία Ντεγλή. Σας συγχαίρω για τη θαυμάσια δουλειά σας, κύριε Λουιαρίκ. Θέλω να επανέλθω σε κάποιες προτάσεις. Δεν θα επανέλθω στις συμβαστικές τροπολογίες. Η, η, πράσινη γενικά είναι ικανοποιημένη. Είμαι ικανοποιημένη επίσης που σήμερα γράφουμε σε ένα κείμενο ότι υπάρχει ανώτατο όριο στις αποδοχές. Λυπάμαι για το εξή μόνο που δεν φτάσαμε σε μια συμφωνία για να προτείνουμε ένα ανώτατο όριο ποσοτικό. Έτσι. Ένα ανώτατο όριο αποδοχών. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα αρχίζει να οριμάζει στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν καλό λοιπόν να προβληματιστούμε το συντομότερο δυνατόν. Εγώ είχα πει ότι θα μπορούσε να είναι το ανώτατο αυτό όριο 44.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 40 φορές ε, το, το μέσο μισθό. Τώρα για το μεταβλητό τμήμα ε, των ε, μισθών. Χαίρομαι για τη θετική άποψη του εισηγητή. Ε, χαίρομαι για την άποψη του εισηγητή που είναι θετική υπέρ των ανθρωπολογιών των πρασίνων, για την ισότητα τη μισθολογική ανδρών και γυναικών και την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Ευχαριστώ. Κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Λεϊάρη που έκανε μια θαυμάσια δουλειά, γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό που έκανε. Για να επιτευχθούν συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες ε, είναι πολύ καλές, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι σημαντική γιατί έλαβε υπόψη δύο απαιτήσει. οι οποίες δεν είναι εύκολο να εξορροπηθούν και στην πολιτική συζήτηση ακόμα. Η πρώτη απέτηση είναι να εισαγάγουμε και να απαιτήσουμε μετά στις συμπεριφορές να δούμε το γενικό επίπεδο των απολαβών των εργαζομένων και τις ευθύνες που ζητάμε από τους ανθρώπους που, που τους δίνουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτούς τους μισθούς. Έπειτα, η άλλη απέτηση είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια στον τρόπο που καθορίζονται οι μισθοί. η διαφάνεια θα μας βοηθήσει στο να υπάρχουν καλές πρακτικές, ε, συνεκτικές ε, δράσεις ε, από τις επιχειρήσεις και θα δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους να μην επωφεληθούν από διάφορες ευκαιρίες που βρίσκουν στην εργασία τους με αήθη τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε κανόνες με τους οποίους θα πορευτούμε για να ξεπεράσουμε την κατάσταση που μας κληροδοτήθηκε. Ε, που δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει από τα πολυάριθμα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα ε, των τραπεζών, αλλά και των υπηρεσιών και της βιομηχανίας. Είναι ένα γενικό πρόβλημα. Πρέπει να δούμε η δραστηριότητα που υπάρχει, οι ευθύνε που αναλαμβάνονται και το επίπεδο αναγνώριση των ευθυνών μέσω των μισθών. Γιατί ο στόχος μας ποιος είναι. Να σπάσει αυτή η ιδέα ότι θα πρέπει να δίνουμε, να δίνουμε ας πούμε μεγάλα κέρδη σε αυτούς που παίρνουν μεγάλα ρίσκα. θα πρέπει να μπορούμε να να δίνουμε, να προωθούμε και συμπεριφορές από πλευράς των εργαζομένων. Δεν θα πρέπει το σύστημα να γίνει άκαμπτο. Οι θετικές συμπεριφορές δεν εξασφαλίζονται μέσω από, μέσα από, τις, μέσα από τους πολιτισμούς. Θα πρέπει να υπάρχει και πειθός και κάποια όρια βέβαια ε, για να προωθήσουμε τις συνεπείς ε, συμπεριφορές. Και νομίζω ότι η στάση του κ. Λιέρη ήταν ακριβώς αυτή. Θέλει κάτι τέτοιο να προωθήσει. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Αλλά νομίζω ότι το σημείο το οποίο, στο οποίο έχουμε φτάσει ε, είναι αρκετά ικανοποιητικό και πρέπει νομίζω να συνταχθούμε όλοι γύρω από αυτό. Ευχαριστώ κύριος Κρότσμαν και μετά η κυρία Πασκάλ Μπρούνι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Μάισνερ βρίσκεται στη Ουάσιγκτον και απατά την επιτροπή σας με μια άλλη αντιπροσωπεία και μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω εδώ. Η κυρία Μάισνερ έχει τονίσει ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πρέπει να υπάρξει και μια μεγαλύτερη αντιμετώπιση των ηθικών θεμάτων που υπάρχουν, αλλά χωρίς υπερβολικές ε, επιβολές κυρώσεων ή περιορισμού. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια υπερβολικά ε, διευθυντική αντιμετώπιση, θα πρέπει να διατηρηθεί η περιορισμου δεν πρεπει λοιπον να υπαρξει μια υπερβολικα διευθυντικη αντιμετωπιση θα πρεπει να διατηρηθει η αρχη της επικορικότητας. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για να ρυθμίσουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Έχουμε πολύ διαφορετικές ε, δομές στα κράτη-μέλη, είναι διαφορετική κατάσταση των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων, επομένως η πολιτική δεν μπορεί να είναι ενιαία. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρουμε πάντα σαν βάση τις ε, υπέρογγες και αστρονομικές ε, αμοιβέ των στελεχών στις ΗΠΑ. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες ισχύουν μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ότι η συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει από τη δική μας πλευρά δεν είναι απλώς να ζητήσουμε να υπάρξει μια ανάληψη ευθυνών των επιχειρηματιών, αλλά να είναι σαφές ότι οι αμοιβέ στο μέλλον θα πρέπει να καθορίζονται από τους μετόχους, οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν και αυτοί την ευθύνη για την λειτουργία μιας επιχείρησης. Γιατί αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το κεφάλαιο στην ιδιοκτησία τους και επομένω την πραγματική ευθύνη για τη σωστή του διαχείριση. Εγώ συμφωνώ επίσης με τις προτάσεις του κυρίου Μπαλτασάρ, η κυρία Μάισνερ, υποστηρίζει επίσης υπέρ των πολλών ε, συμβαστικών τροπολογιών οι οποίες έχουν κατατεθεί και αυτά ήθελα να σας πω εκ μέρους της. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Πασκάλ Γκρίνι, Έλμα, μετά. Ναι, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ιδιαίτερα με ενδιέφερε η γνωμοδότηση αυτού του κυρίου Λεγιάρικ μετά από τη δημοσιομενική αυτή κρίση, την οικονομική, την κοινωνική, που προέρχεται από μια κακή διαχείριση από τις τράπεζες, θα πρέπει να δούμε από πιο κοντά τι γίνεται με τα κεφάλαια, πώς τα διαχειρίζονται και για τις αποδοχές, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι κάτι σαν όσον την αναλογία τους με ευθύνη να βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Οι αποδοχές αυτές ε, χρειάζονται να μπορούν ε, να τις καταλάβουν, να τις αποδεχτούν και οι πολίτες μας. Ε, δεν είμαι υπέρ του να υπάρξει ένα ανώτατο όριο, γιατί τότε θα βάλουμε φράγματα. Μπορούμε να θέσουμε ανάμερα με, κριτήρια, με κύκλους εργασιών και άλλα παραμία. Δεν ξέρω πώς τα που θα οδεύσω μετά, αλλά δύσκολο θα είναι. Και οι συνάδελφοι πριν να δουν τώρα ποιοι είναι υπεύθυνοι των τραπεζών που αναλαμβάνουν κινδύνους. Πάρα πολλή δουλειά να, να κάνουν. Η συνάδελφος λοιπόν ε, ε, είδε πρώτα την επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου που έχουν αποδοχές που μπορούν να μας βάλουν σε σκέψεις. Και θα πρέπει να δούμε και το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα σε αυτή την έκθεση. Το σύνολο της έκθεσης αυτής ε, για αυτά τα υποχρεωτικά ποσοστά δεν μπορώ να τα υπερψηφίσω, αλλά όχι στην 16, μάλλον ναι στην 16 θα την υπερψηφίσω, αντιστοιχεί σε αυτό που εγώ επιθυμώ, δηλαδή σε αυτά τα μέτρα δεσμευτικού χαρακτήρα, χωρίς όμως να βάλουμε ανώτατα όρια. Αυτά θα ήθελα να πω και να υποστηρίξω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και η πρόεδρος Έλμερτ και μετά Τόμας Μαν. Uh, Δεν κατάλαβα ότι μιλούσατε για μένα κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Παρακολουθώ. Διακόπτη Πρόεδρος. Ναι, ναι, θα... Θα μιλήσω στα αγγλικά, δεν σας πειράζει, κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Θα έλεγα ότι είμαι ενευρόντιτος από αυτή τη συζήτηση. Γιατί ξεκίνησα με ένα ερώτημα για τον εαυτό μου. Τι θα πει δεοντολογία. Εγώ έχω μελετήσει, έχω μελετήσει την αγγλική γλώσσα εδώ και 65 χρόνια. Δεν νομίζω ότι την αγγλική γλώσσα δεοντολογικός, deontological. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Όλη η συζήτηση βασίζεται σε μια υπόθεση ότι οι τράπεζες και τα άλλα τα επιστοτικά ιδρύματα είναι απόλυτα υπεύθυνοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ίσως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν φτάνει μονάχα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όλα αυτά τα προβλήματα ξεκίνησαν στην Αμερική με τον πρόεδρο Jimmy Carter και τον διάδοχό του που ουσιαστικά παρότριναν τα ιδρύματα που έδιναν στεγαστικά δάνεια να δώσουν και τις τράπεζες να δώσουν δάνεια σε όλους. Ο Άλαν Γκρίτσπαν κράτησε χαμηλά τα επιτόκια για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τον ακολούθησαν οι ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό οδήγησε σε μια φούσκα σε ό,τι αφορά τις τιμές των ακινήτων. Κάποιοι θεσμικοί φορείς πήραν λανθασμένες αποφάσεις. Δεν φταίνε τα ψάρια που κολυμπάνε στο νερό λοιπόν. Είναι η δουλειά των κρατών να θεσπίζουν μια σωστή νομισματική πολιτική και λογικά επιτόκια και να ρυθμίσουν τις χρηματαγορές. Δεν είναι δουλειά των κρατών όμως ή του Κοινοβουλίου μας ή της Επιτροπής μας να έχουν παρεμβατική νομοθεσία σε σχέση με τα επίπεδα αμοιβών και αποδοχών μέσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εγώ θα έφερα τον κύριο Κρότσπερτ σε κάποια δυσκολία. Ευτυχώς έφυγε γιατί συμφωνώ μαζί τους είναι σωστό αυτό που λέει ότι είναι κάτι που εναπόκειται σε εταιρείε και του μετόχου να το αποφασίσουν αυτό και όχι στην Επιτροπή μα. Δεν είναι δουλειά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη δική μα Επιτροπή να καθορίσει του φορολογικού συντελεστέ. Άκουσα τη συζήτηση για το πώ θα πρέπει να φορολογείται το εισόδημα των στελεχών. Όλη αυτή η ιδέα των υποθηκευμένων φόρων έχει αναφερθεί χωρί να υπάρχει παραμικρή αιτιολόγηση για κάτι τέτοιο. Εμεί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Επιτροπή μα μπορούμε να αποφασίσουμε πώς θα πρέπει να συλλέγονται οι φόροι, σε ποιο επίπεδο και πώς θα πρέπει να δαπανούνται. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι κάτι μεταξύ του σκανδαλωδού και του παράλογου. Έχω τεράστια δυσκολία λοιπόν να υποστηρίξω μια από αυτέ τι προτάσει που περιέχεται σε αυτή την έκθεση, ακόμα και τι συμβαστικές τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε αγαπητέ. Δίπλα μου είναι ε, ειδικό ε, στα ελληνικά μάλιστα τα γνωρίζει πολύ καλά που λέει ότι από τα αρχαία ελληνικά έρχεται αυτό το δεοντολογικό και να σας διαβάσω και τον ορισμό που έχω στο λεξικό μου επίσης καθενονισμοί επαγγελματικοί, επίσης ιατρική διοντολογία και το καθήκον του ιατρού που έχει να κάνει και με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα νομίζω ότι είναι και στα δημοσιονομικά κλπ. Τόμας Μαν και Μωράν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ μπορώ να σας ονομήσω να σε ονομάσω Madame La Présidente και όχι απλώς Madame Le Président. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το άτομό σας. Δυστυχώς ο κύριος Κρότσμπερκ έφυγε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήθελε να ακούσει τη συνεδρίαση και τη συζήτηση. Πρέπει να πάει σε μια άλλη επιτροπή όπου θα έπρεπε να συμμετάσχει στη συζήτηση. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεγάλη ευθύνη και οι οποίε είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Γνωρίζω τα άτομα αυτά τα οποία βρίσκονται σε αυτέ τι επιχειρήσει και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ υπάρχουν άλλε επιχειρήσει που κάνουν ό,τι θέλουν. Συνεχίζουν τη δουλειά του και παίρνουν τα πριν του. Επομένω, θα πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι και ο ρόλο των επιχειρήσεων για τον κοινωνικό πλαίσιο των κοινωνιών μα. Έτσι πρέπει να δούμε τα θέματα των αποδοχών είχα την ευκαιρία να συζητήσω με άτομα τα οποία είναι υπεύθυνοι για μεγάλες τράπεζες. Τους είπα είναι δικαιολογημένα τα μπόνους σας, τα πρέμ σας. Είπανε ότι εμείς οι επιχειρήσεις μας στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη παίρνουμε μπόνους μόνο όταν έχουμε θετικά αποτελέσματα για τέσσερα χρόνια τουλάχιστον. Όχι γιατί αγοράζουμε κάτι, πουλάμε και αμέσως έχουμε κάνει κέρδος. Επομένως είναι απαραίτητο να τονίσουμε το να υπάρχει διάρκεια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις κερδοφορίες τους, να έχουμε εταίρους οι οποίοι βασίζονται σε αυτό, αυτό είναι κατελείως διαφορετικό, γιατί το να υπάρχει διάρκεια και αηφορία, αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο επίπεδο σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των πριν. Αλλά τώρα, όταν μιλάμε για το ύψος των πριν και των αποδοχών, Αυτό μπορώ να το κατανοήσω αν έχουν πραγματικά μια υπευθυνότητα οι εργαζόμενοι την οποία να την φέρουν σε πέρας. Θα έπρεπε μέσα στα πλαίσια της κρίσης να υπάρξει μια απόφαση να μειώσουν τις αποδοχές τους και τότε όταν βγει κανείς από την κρίση μπορούν να αυξηθούν πάλι οι αποδοχές τους διότι θα έχει εξέλθει η επιχείρησή τους και η οικονομία τους από την κρίση. Αυτό είναι μια ηθική στάση, μια διοντολογική στάση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει τα στελέχη να ξέρουν ότι έχουν και αυτοί μια πραγματική ηθική ευθύνη για να μπορέσουν να συμπεριφερθούν όπως πρέπει μέσα στα πλαίσια μιας κρίσης. Μέσα σε αυτό το πνεύμα εμεί έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που νομίζω ότι εξισορροπούν κάπως καλύτερα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Κυρία Μογά, και Ξανά η κυρία Ντελή δεν συνηθίζεται, αλλά μια και έχουμε χρόνο θα μπορούσαμε να τη δώσουμε το λόγο. Η κυρία Μογά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μέσα σε αυτό το γικαιώνα τον οικονομικό που γνώρισε όλος ο πλανήτης. Σημερίζομαι και αυτά που είπε ο Τόμας Μάν μόλις τώρα και η Πασκάλ Γκουινή πριν από λίγο. Πρέπει να αποφύγουμε να στυλιτεύσουμε ως ληστές και δολοφόνους τους πάντες. Υπάρχουν άνθρωποι που όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο έχουν και ηθική και ιδεοντολογία στις επιχειρήσεις και στις τράπεζες σέβονται τους κανόνες που είναι σαφείς, κατανοητοί από όλους. Βεβαίως, πρέπει να σεβόμαστε αυτούς τους χώρους που είναι πολύ δυναμικοί. Αυτοί δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και οι θέσεις απασχόλησης πληρώνουν τους μισθούς στους εργαζόμενους. Πρέπει να τους αφήσουμε περιθώριο να κινηθούν. Να, υπάρχει μια πλαισίωση, αλλά πρέπει να υπάρχουν, και βέβαια πρέπει να υπάρχουν κανόνες ε, δεοντολογίας, αλλά δεν θα πρέπει να φρενάρουμε τις δραστηριότητές τους με υπερβολικά επιτακτικές ρυθμίσεις στους μισθούς που θα ε, δημιουργούσαν μια τροχοπέδη στις οικονομικές δραστηριότητες. Ε, λίγοι κανόνες είναι καλοί, αλλά οι υπερβολικοί κανόνες είναι αντίθετοι στα συλλογικά μας συμφέροντα. Τώρα, για την τροπολογία 16, εγώ προσωπικά έχω ακριβώς την ίδια θέση με την κυρία Γκοϊνή για τους ίδιους ακριβώς λόγους που σε εξέθεσε εκείνη. Κυρία Ντελή, μέσα σε δύο χρόνια αυτή η οικονομική κρίση κόστισε τη δουλειά πάνω σε 10 εκατομμύρια εργαζόμενους. Δηλαδή έμειναν άνεργοι αυτοί οι άνθρωποι. Και παράλληλα έχουμε αήθιες πρακτικές, μπόνους παντού στη ΣΥΤΗ που έχουν αυξηθεί κατά 50% το 2009 σε σχέση με το 2008 ε, φτάνουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, στο Παρίσι έχουμε μπόνους ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και εσείς μιλάτε για διοντολογία παρ' όλα αυτά. Προηγουμένω μου είπατε για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Να υπενθυμίσω ότι σε εποχή κρίση το, το 42 Ρούσβελτ είχε μιλήσει για το ανώτατο α, μισθό για να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Το θέμα της διοντολογία σημαίνει κοινωνική ευθύνη. Και αυτό το σχέδιο αυτό το σχέδιο νομοθετήματος αφορά ε, τις επιχειρήσεις, αφορά τους εργαζόμενους. Ε, ας αφήσουμε κατά μέρος τους ε, ποδοσφαιριστές. Ο κ. Κλάρκ. Ας αφήσουμε τώρα την ορολογία και τη διοντολογία. Γιατί... Βάσει της αιτιολογικής σκέψης α, αναφέρεται το, η διοντολογία όπως η διαφάνεια στη διαχείριση του κινδύνου, ή η άσκηση των δικαιωμάτων των... Ε, Μπορώ να σας διακόψω, λέει η πρόεδρος. Διαβάζετε την έκθεση, λένε. Ναι. Σας μιλάω στα αγγλικά, δεν χρειαζόσαστε αυτά τα ακουστικά. Μα δεν σας ακούω, κυρία μου, λέει ο μιλητής. Διαβάζετε την έκθεση, λένε, ναι, που είναι η έκθεση, λένε, στην κυρία Επιτροπή. Δεν είναι η έκθεση όμως του κυρίου Λεγιαρίκ. Μα φαίνεται ότι εξηγεί αυτή η έκθεση το τι ακριβώς είναι η δεοντολογία που είναι αυτό το οποίο συζητούμε. Μήπως μπορώ να συνεχίσω. Δεδομένου του ότι η δεοντολογία λοιπόν παίζει κάποιο ρόλο, είναι σωστό οι επιχειρήσεις να παίρνουν συμβουλές από αυτούς που έχουν αναλύσει, όπως λέει η έκθεση αυτή, τα θέματα και έχουν καταθέσει σε κάποιες προτάσεις αλλά δεν μπορείτε να τους διατάξετε να ακολουθήσουν τις συμβουλές αυτές. Δεν μπορείτε να πείτε στις επιχειρήσεις πώς θα οργανωθούν. Δεν μπορεί η Επιτροπή μας να φτιάξει ένα πλαίσιο που λέει στους επιχειρηματίες πώς θα δραστηριοποιηθούν και πώς θα λειτουργήσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το απορρίπτω διαρρήδην. Να υπάρχουν συμβουλές, ναι. Να υπάρχουν υποχρεώσεις, όχι. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θα επιθυμούσε το λόγο. Α, κυρία μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία προσθήκη, μία παρατήρηση μου μορφή προστίκης θα ήθελα να κάνω, στεκόμενη σε ένα σημείο που εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή την πλευρά της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, δηλαδή να μπορούν και οι γυναίκες να λαμβάνονται υπόψη πλήρως μέσα στα πλαίσια αυτής της προβληματικής που εξετάζουμε. Η Κομισιό λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της για να προωθήσει την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Ανεξάρτητα λοιπόν από όλες τις άλλες πτυχές της χρηματοοικονομικής κρίσης, αυτό είναι μια πτυχή η οποία πρέπει και αυτή να ληφθεί υπόψη η παρουσία των γυναικών, δηλαδή σε ηγετικές θέσεις. Ε, Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θα επιθυμούσε να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Κύριος Ντερόσα. Ευχαριστώ. Ε, άκουσα αυτή τη συζήτηση για τη διοντολογία και για το ότι δεν είναι αγγλική λέξη. Κύριε Χέλμερ, η αγγλική γλώσσα, παρότι είναι Ιρλανδός, είναι και δική μου μητρική γλώσσα. Μην ξεχνάτε ότι το 50% των αγγλικών λέξεων που υπάρχουν δηλαδή στο αγγλικό ε, λεξικό προέρχονται από τα γαλλικά. Αλλά και κάποιες κοινέ ρίζες με τα ελληνικά έχουν τα γαλλικά. γλώσσες ε, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς εκεί ανήκουν. Ε. Και αρκετές είναι λατινικές από τις γλώσσες μας. Τα γύρω από τη Μεσόγειο. Βλέπουμε λοιπόν τις ρίζες του πληθυσμού μας, του πολιτισμού μας ε, κάπου εκεί, γύρω από τη Μεσόγειο. Αυτή την εποχή τουλάχιστον χρησιμεύει να τα υπενθυμίζουμε. Κάποιος άλλος που θα επιθυμούσε το λόγο. Όχι κανείς. Έχει και πάλι, ο εισηγητής μας το λόγο. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που συμμετείχατε στην συζήτηση αυτή. Για τρεις μικροπαρατηρήσεις να κάνω. Για το ερώτημα που τέθηκε για τις διάφορες αυτές ε, επιχείρησεις. Ε, το καθένα από αυτά δεν ε, σημαίνει και ένας επικεφαλής και δεν είναι ότι παίρνει περισσότερα χρήματα από ότι οι υπάλληλοι τα ίδια λοιπόν δεν τους αφορά. Κάτι που ρωτούν τώρα για τον νομοθετή κανείς ή όχι πάνω σε αυτό. Διεξάγεται μια συζήτηση, προσφέρουμε μια γνωμοδότηση το τι θέλουμε να το ξέρουμε. Εκλεγμένα από το λαό για την όλη διοίκηση αυτής της οντότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν θα πρέπει να φέρουμε σε αυτό το επίπεδο τη συζήτηση. Εάν θέλει κανείς να πει ότι χρειάζεται να οργανώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να νομοθετήσει, είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία αυτή ακριβώ Είμαστε εκπρόσωποι εμεί. Διαφορετικά ο καθένα κάτι ό,τι θέλει. Αλλά τι διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Κάποιο έκανε μια παρατήρηση. Σύμφωνα με την παρατήρηση αυτή υπάρχει μια πρόσβαση συνεχή. Τι βλέπω εδώ, ότι θα αυξηθεί ένα φόρο, θα είναι φόροι. Ο ΦΠΑ αυξάνεται για του Έλληνε, αλλά όχι επιπλέον φόροι σε αυτούς τους φόρους που αφορούν την κατάσταση αυτή. Μια άλλη παρατήρηση ακόμα. Εμείς εδώ αυτά που συζητούμε και αλλού άλλους χώρους ε, συζητούνται και μάλιστα με περισσότερο ενδιαφέρον ε, στο G20 ας πούμε δύο, φορά, δύο φορές ε, και από τις Ευρωπαϊκές Αρχές και στο Συμβούλιο Οικονομικών διεξήχθησή το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βλέπουν όλοι πολύ καλά λοιπόν ότι ναι, απαιτούνται αποφάσεις νομοθετικού χαρακτήρα. Διαφορετικά, επαναλαμβάνω, θα επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Να το διαλύσουμε μετά. Όχι, ε, δεν θα ήθελα το ε, προτείνω αυτό. Είμαι κατά της νόμου της ζούγκλας ε, και τα θύματα είναι τα ίδια αυτοί που έχουν την εργασία τους ή την σύνταξή τους για να ζήσουν. Πάντως σας ευχαριστώ για όσα είπατε, ήταν επικοδομητικά, θετικά. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Νομοδότηση λοιπόν, θα το δούμε αυτό και στην ψηφοφορία αύριο. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο, το 7. Το λόγο έχει ο συνάδελφό μας Σέρτζιο Γκαϊτάνο Κοφεράτη για την ε, Επιτροπή Οικονομικών για την ανάκαμψη της οικονομίας μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Κύριε Σεγητά, έχετε το λόγο. Ο κύριος λοιπόν Κοφερατή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω εγώ όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι σχολίασαν το κείμενο το οποίο τους είχα δώσει Στη συνέχεια δε κατέθεσαν τροπολογία στα πλαίσια μιας ευρείας συνεργασίας, κάτι που ιδιαίτερα με χαροποίησε. Να ομολογήσω ότι το μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών που πήρα στα χέρια μου και από την Πρόεδρο και των υπολείπων συναδέλφων, οι τροπολογίες αυτές είχαν σαν στόχο να διευκρινίσουν, να εμπλουτίσουν τον αρχικό στόχο στα πλαίσια αυτού του οικοδηματικού πνεύματος. Και έτσι μπορέσαμε να συντάξουμε και ορισμένα κείμενα. που συμφωνήσαμε με τα κύρια στοιχεία από αυτές τις τροπολογίες, έτσι έχουμε στα χέρια μας λύσεις για μία πλατιά σύγκληση. η μοναδική συνάδελφος που θεωρώ ότι οι τροπόλογοι της ε, δεν μπορούν να γίνουν από μένα δεκτές είναι η κυρία Φιγκερέιντο. Η άποψή της είναι διαφορετική για τον πυρήνα του θέματος που εξετάζουμε. Για να δούμε λοιπόν. Εντάξει, όλα αυτά γίνονται. Γιατί όχι. Μέρο ε, ενός ε, διαρθρωμένου καλά σχεδίου, αλλά σίγουρα εναλλακτικού σε σχέση τουλάχιστον με το κείμενο το οποίο οι υπόλοιποι σχολίασαν και κατέθεσαν τις τροπολογίες στη συνέχεια. Γι' αυτό δεν μπορώ να τις δεχτώ, τις τροπολογίες της κύριας Φιγκερέιντο. Τις σέβομαι βέβαια, τις τροπολογίες αυτές. Τις υπόλοιπες τις επεξεργαστήκαμε και με συμβιβαστικές λύσεις που κατά την απόψή μου ήταν αποτελεσματικές, θετικές. Να σας μιλήσω για μία πτυχή από όλα αυτά. Έχει να κάνει με την συζήτηση που διεξήχθη και που σε δύο συμβαστικές λύσεις δεν επέτρεψε τη σύγκληση που πίστεψα θα μπορούσαμε να πετύχουμε στην αρχή τουλάχιστον το πίστεψα αυτό. Εδώ σε τι αναφέρομαι ειδικά. Συμβαστική λύση γάμα. Σι λατινικό. Και το πέντε το ε το λατινικό. Δεν πετύχαμε λοιπόν τη σύγκληση όπως το ευχόμουν. Το ίδιο και για την γάμα και για την ΕΨΙΛΟΝ τροπολογία. Συγχωρήστε με λοιπόν θα κάνω χρήση του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου για να επανέλθω σε αυτό που δεν έπεισε τους συναδέλφους. Την συνάδελφο κυρία Γεροζέλσκια. Σχετικά με τις αποδοχές για το πώς κανείς μπορεί να τις υπερασπιστεί. Πριν από λίγο το είδαμε το θέμα αυτό. Το εξετάσαμε να επιμείνω πάνω στο κείμενο των δύο συμβαστικών λύσεων. Και για ένα προφανή λόγο. Πάντα είναι πολύ σημαντικό και τώρα ακόμα περισσότερο σε παρόμοια τρομερή κρίση όπως αυτή που διανύουμε. Το να έχουμε στα χέρια μας μέσα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη ρύθμιση της κατανομής του πλούτου που παράγεται και εργαλεία φορολογικά αλλά και μέσω συμφωνιών, συλλογικών συμβάσεων κλπ. Εκεί που υπάρχουν, που ισχύουν αυτές οι συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους. Και ήττος και για το welfare, για τρευμάρια αυτά τα χρήματα για να μπορεί κανένας να ζήσει αξιοπρεπώς Λοιπόν, δεν θέλεις να λάβω υπόψη μου αυτό τα δεσμευτικά για τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει κανείς να υπερασπιστεί την ζωή των ε, προσώπων των διαφορών ατόμων και υπερασπιζόμενες τις αποδοχές τους, γιατί τα μέσα ποικίλουν ιδιαίτερα από τη μία χώρα στην άλλη. Αλλά αυτή η αρχή, αυτή είναι η έννοια αυτό που έπρεπε να υπερασπιστούμε σε όλους είναι μια αξιοπρεπή ζωή μέσω ενεργειών που κυρίως προέρχονται από πλευράς κυβερνήσεων και μας ε, οδηγούν προς την κοινωνική προστασία και άλλες ενέργειες στα πλαίσια συλλογικών συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό δε μπορούμε και να υπερασπιστούμε και το πώς ζουν υλικά και τις συντάξεις και και τις αποδοχές τους οι αποδοχές, κάτι που δεν εξετάζουμε εδώ, αλλά στα πλαίσια αυτής της περίληψης που προσπάθησα να προτείνω, θα έπρεπε πάντα να ανταποκρίνεται και στον επαγγελματικό χαρακτήρα του εργαζόμενου ατόμου. Πώς η ποσότητα εργασίας παράγει, που έχει να κάνει και σε πόσο χρόνο μέσα το κάνει αυτό. Και για την παραγωγικότητά του επίσης. Και αυτό μέσω της συγκεκριμένης εργασίας του εν λόγω ατόμου. Μια ίση σχέση λοιπόν ανάμεσα στην παροχή υπηρεσία, στην εργασία, στο αποτέλεσμα, στην αποδοχή. όλα αυτά μπορούμε κανείς να τα συμμεριστούμε, μπορούμε να τα συμμεριστούμε. Δεν ε, αποκλείει την κατάλληλη σχέση ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο, αλλά δείχνει μια κάποια παρότριση, ένα κάποιο κριτήριο προσφέρει για μια αποτελεσματική συμπεριφορά, για μια σωστή πρακτική. Αυτό, στα όσα πρότεινα εγώ, στα κείμενα αυτών συμβαστικών λύσεων, ανταποκρίνονται σε αυτή τη λογική, λογική και όχι έτσι κατευθυντήριες γραμμές και δεσμεύσεις. Σε αυτές δεν πιστεύω και λόγω πολιτικής ε, φιλοσοφίας και ορισμένα που επαγγελματικά διδάχτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτά θα αρκεστώ. Γιατί οι τροπολογίες, οι υπόλοιπες εκτός της κυρίας Φιγκερέιντο, όπως είπα, οι υπόλοιπε στο σύνολο του Σελίου περίπου τις αποδέχομαι γιατί έχουν ε, μια θετική χρειά την οποία και εκτίμησα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας λέω κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κύριε Κοφεράτη για τη θαυμάσια δουλειά σας. Διατρέχοντας τις προτάσεις και τις συμβαστικές τροπολογίες, ε, συνειδητοποίησα ότι αυτή η έκθεση, ε, η τροποποιηθήσα έκθεση, αυτό που κάνει είναι ότι λέει, κοιτάξτε, από τη μία έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ρυθμίσουν τα αφρολογικά τους. Αυτό σημαίνει μείωση και των δαπανών από τη μία, αλλά από την άλλη λέμε «Α, δεν μπορείτε να μειώσετε τις δαπάνες εδώ, εκεί και παρακεί». Επομένως, τελικά πώς συνεισφέρουμε δηλαδή για να επιληθούν τα οικονομικά προβλήματα, γιατί καθορίσουμε δύο στόχου που είναι επιθυμητοί, αλλά είναι ασύμβατοι μεταξύ Ε, συμφωνώ ότι οι περισσότερε κυβερνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μειώσουν τι δαπάνε του για να βελτιώσουν τα δημοσιονομικά του, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι πρέπει να μειώσετε τι δαπάνε για να βελτιώσετε τα δημοσιονομικά σα και μετά να δίνουμε ένα ολόκληρο κατάλογο τομέων όπου δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να κόψουν τι δαπάνε. Αυτό ε, τι συνέπεια έχει τελικά. Δεν μπορεί να κόψετε καμία δαπάνη Κοιτάξτε, ας αποφασίσουμε. Ή θέλουμε ή δεν θέλουμε να κόψουμε τις δαπάνες. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι καθώς εξετάζουμε αυτές τις τροπολογίες, οι οποίες απλώς προσθέτουν νέους στόχους, στην πραγματικότητα φτιάχνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπου τα κράτη-μέλη, συγγνώμη, οι βουλευτές μάλλον, και κυρίω οι αριστεροί βουλευτέ μπορούν να βάλουν όλε τι μπαλίτσε, α πούμε, στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που επιθυμούν. Ούτω ή άλλω αυτά θα μπορούσαμε να τα ζητήσουμε οποτεδήποτε. Αλλά τα ζητάμε σε μια εποχή όπου τα μέσα, τα φορολογικά μέσα των κρατών μελών για να υλοποιήσουν αυτού του στόχου είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Επομένω, καταλήγω λέγοντα ότι δεν καταλαβαίνω πώ αυτή η έκθεση, έτσι όπω έχει ή όπω μπορεί να τροποποιηθεί, πώ μπορεί να συνεισφέρει τελικά. Πώ μπορεί να συνεισφέρει στα προβλήματα που έχουμε εμεί και οι Ευρωπαίοι πολίτε. Σας ευχαριστώ αγαπητέ για τη βοήθεια αυτή. Κύριος Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σταθώ σε τρία θέματα μέσα σε αυτό το θέμα. Εγώ είμαι ευγνώμων στον εισηγητή που λέει ότι στο σημείο 9 ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στο ασφαλιστικό σύστημα και να μπορέσει να διευρυνθεί η βάση χρηματοδότησης αυτού του ασφαλιστικού συστήματος. Θα ήθελα να πω εδώ ότι αυτό δεν είναι μονάχα ένα σύστημα το οποίο υποστηρίζει τον κοινωνικό ιστό, την υγειονομική περίθαλψη κτλ. Θα πρέπει αυτό όμως να το συνδέσουμε και με την παροχή συντάξεων, με το συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο πρέπει να συνδεθεί με αυτή την προβληματική. Στο σημείο 10 θα ήθελα ο εισηγητής να έχει μια σαφέστερη μνήα αυτού το οποίο είπε πρόσφατα ο Επίτροπος Αλμούνια ενώπιον της Επιτροπής μας και το οποίο έχει διατυπωθεί ήδη από την Επιτροπή ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχει φτάσει η ηλικία συνταξιοδότηση σε πολλές χώρες στα 67 και ότι σε πολλές άλλες χώρες είναι απαραίτητο να ανέλθει η ηλικία συνταξιοδότησης ώστε να είναι διατηρήσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν ο εισηγητής να έχει λάβει υπόψη αυτή την προβληματική σε σχέση με την ε, ηλικία συνταξιοδότησης. Αναφέρθηκε η τροπολογία της κυρίας Φιγκερέδο, της συναδέλφου μου, η οποία επεκρίνει εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτή η κριτική δεν είναι δικαιολογημένη, νομίζω ότι είναι και λανθασμένη εξάλλου. Στην τροπολογία 9 αναφέρεται εκπεφρασμένα η διατύπωση της κυρίας Φιγκερέδο που λέει ότι πρέπει να υπάρξει η ανάπτυξη ποιοτικών και ε, υψηλής ποιότητας εργασιών. Νομίζω ότι η Επιτροπή της ε, απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ενώπιον μιας αναδυόμενης παγκόσμιας ένδυας είναι απαραίτητο να υπάρξει μια καλύτερη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος ώστε να αντιμετωπιστεί και η ένδυα η οποία υπάρχει. Θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη το ότι εφέτος ήταν το έτος ε, κατά της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού να συμπεριλάβει και αυτή την μνήα στην έκθεσή του. Merci. Ε, Σας ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ. Ε, καλύτερα να λέτε Ντάνα με το μικρό, είναι πολύ πιο εύκολο. Ε. Το επώνυμό μου είναι πολύ δύσκολο να το προφέρετε σωστά. Ντάνα καλύτερα. Ε, έχετε το λόγο, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην έκθεση Κοφεράτη, στην γνωμοδότηση μάλλον Κοφεράτη, σε σχέση με την έκθεση της Κομισιόν για την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, αυτό που δεν υπάρχει είναι η ρευστότητα των δημοσίων οικονομικών. Δεν μιλάμε καθόλου για το τι είναι αυτό που παράγει την οικονομική ανάπτυξη. Δεν μιλάμε για την γύρανση του πληθυσμού και δεν μιλάμε για την παράταση της επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή του, χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Γι' αυτό πρότεινα τρεις τροπολογίες. Παραδείγματο χάρη για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων σύνταξη, μιλάτε για δύο πυλώνε για τη χρηματοδότηση του συστήματο, ενώ εγώ προτείνω τρει πυλώνε, τα, το δημόσιο, τα δημόσια κονδύλι, κονδύλια, ε, τι συνεισφορέ από, τις, από του μισθού και τι συνεισφορέ από τις αγορέ. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των συντάξεων. Ένα άλλο θέμα αφορά την ε, μετανάστευση. Για σας είναι θετικό για να διορθωθούν τα δημογραφικά προβλήματα των κρατών μελών. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους ανθρώπινους πόρους, να τους εμπλουτίσουμε και να μην ε, προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις μόνο και μόνο στην μετανάστευση. Να τονίσω και ένα άλλο αρκετά σημαντικό σημείο. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των ε, δαπανών από το δημόσιο κορβανά θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός των σημερινών ε, δεσμεύσεων και των μελλοντικών δεσμεύσεων, κυρίως οι δεσμεύσεις σε σχέση με τα κοινωνικά θέματα. Να, θα πρέπει να υλοποιούνται αυτές οι δεσμεύσεις. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας όλους. Ο κύριος Κοφεράτη έχει συντάξει έξι συμβαστικές τροπολογίες. Όλες αυτές ε, οι συμβαστικές ε, τροπολογίες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με τη δική μας για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες α, β και δ, αυτές τις συμμεριζόμαστε. Αλλά για τις υπόλοιπες CF, CE και F, Αυτές ε, κινούνται σε κάποιο βαθμό προς ε, διαφορετική κατεύθυνση από του ΕΛΚ. Να σας εξηγήσω γιατί σε για ΣΥ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αναφορά στις φορολογικές πολιτικές για την προστασία των μισθών, των συντάξεων και των επιδομάτων ανεργίας. Σας είπατε μάλλον ότι δεν καταλαβαίνετε γιατί δεν συμφωνούμε. Θα το εξηγήσω σε λίγο. Για την τροπολογία Ε, ε, δεν συμφωνούμε με την αναφορά στην υποστήριξη δίκαιων απολαβών. Γιατί καλό θα ήταν να έχουμε ορισμούς για αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες. Για την ε, F, η αναφορά στις, ε, στα δημοσιονομικά και στις οικονομικές πολιτικές, που βασίζεται στην αναδιανομή του εθνικού πλούτου, αυτό είναι απαράδεκτο. Η κρίση δείχνει ότι στις χώρες όπου έγιναν αλλαγές και στα συστήματα συντάξεων, οι χώρες αυτές ε, περνάνε πιο εύκολα από την οικονομική κρίση και διέρχονται αυτής με μεγαλύτερη ευκολία. Θα πρέπει να αναζητήσουμε μία λύση που δεν θα μειώνει το επίπεδο των συντάξεων και δεν θα δυναμητίζει το επίπεδο ζωής. Το να υπάρξει πάγωμα θα ήταν πολύ κακό. Πάγωμα των συντάξεων και των μισθών θα ήταν πάρα πολύ κακό. Γι' αυτό λοιπόν δεν συμφωνούμε με αυτές τις τρεις τροπολογίες C, και F. Ε, Κυρία μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω τον κύριο Κομφεράτη για την γνωμοδότηση την οποία έχει συντάξει. Πρέπει να πω ότι 99% αυτού του εγγράφου είναι πολύ καλά συντεταγμένο και ισορροπημένο και η πολιτική μας ομάδα θα υποστηρίξει τη γνωμοδότηση του κυρίου Κομφεράτη. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε την πολιτική οικονομικής ανάκαμψης με μέτρα κατά της ανεργίας. Είναι σαφές ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας με ποιότητα θα αυξήσει και την αποδοτικότητα των επενδύσεων. Οι διατυπώσεις αυτής της χρωμοδότησης που αναφέρονται στη φορολογική πολιτική έχουν ένα λογικό χαρακτήρα. Για τις συμβαστικές τροπολογίες δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα γιατί αύριο θα γίνει ψηφοφορία και θα δούμε τι θα προκύψει. Έχω ένα ερώτημα. Η κυρία Λισλίν έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες και δεν έχω κατανοήσει γιατί ο κύριος Κομφεράτη δεν έχει δεχτεί την τροπολογία 4 γιατί είναι πολύ παραπλήσια με τη δική του τροπολογία, με τις ιδέες που έχει διατυπώσει ο ίδιος και η τροπολογία 4 ουσιαστικά διαλευκάνει ακόμα περισσότερο τις ιδέες του κ. Κομφεράτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει. Πρόεδρος, μήπως κάποιος άλλος τώρα επιθυμεί να λάβει το λόγο. Δεν βλέπω. Εκπρόσωπος Επιτροπής παρόν εδώ. Ο κ. Κοντέζο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω τη γνωμοδότηση που προετοίμασε ο κύριος Κομφεράτη που θεωρούμε ότι δίνει μερικά πολύ εύστοχα μηνύματα στον χώρο της πολιτικής. Δυστυχώς δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να δω τις συμβαστικές τροπολογίες μπορώ να πω κάτι για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί καταρχήν πριν από τις συμβαστικές τροπολογίες. Καλωσορίζουμε την εστίαση του εισηγητή για την επίτευξη μιας ισορροπίας και της παγίωσης των δημοσίων οικονομικών, ιδίως στο φως της δημογραφικής γύρανσης και αυτό καταγράφεται και σε ορισμένε από τι τροπολογίε που έχει καταθέσει ο κ. Κοφεράτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίση, από την συζήτηση διεφάνει ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προσοχή που δίδεται στις αποδοχές των εργαζομένων. Και το ερώτημα είναι ποια είναι η πολιτική η οποία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις βραχυπρόθεσμες ελλείψεις ισορροπίας και ανισότητες και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι οι αποδοχές των εργαζομένων θα πρέπει να λάβουν υπόψη την εξέλιξη στην παραγωγικότητα και επομένως όπως αναφέρεται και από τον κύριο Κοφεράτη θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη από την πλευρά της από τη δική μας πλευρά, την Κομισιόν, γιατί σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει παραλληλία παραγωγικότητας και αποδοχών. Φυσικά δεν μπορούμε να δεχτούμε όλα αυτά τα οποία έχουν προταθεί εναντίον του συμφώνου για την σταθερότητα που είναι πολύ χρήσιμο αυτό το σύμφωνο για τον συντονισμό των πολιτικών. Αυτό θέλω να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητή έχει τον λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Κρίμα που έφυγε ο κύριος Χέλμερ. Θέλω να τον καθησυχάσω όμως. Εγώ δεν σκέφτηκα να φτιάξω σε καμία περίπτωση ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο για να βάζει ο καθένα τον μπαλάκι του. Γιατί στο κάτω-κάτω στη δική μου κουλτούρα, εμεί δεν έχουμε το δέντρο, αλλά έχουμε τη φάτνη. Ε, με δώρα. Ε, και τους μάγους που πηγαίνουν για να αποτίσουν φορό τιμής στο νεογέννητο Ιησού. Ε, έτσι λοιπόν, ε, ξέρετε ότι στη Φάτνη επιλέγουμε. Επιλέγουμε τις μορφές. Ε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό η Φάτνη από το δέντρο. Και λοιπόν εγώ με αυτή τη λογική έφτιαξα την έκθεσή μου, την ε, με την προσπάθεια να προωθήσω τις επιλογές. Προσπάθησα να αναφερθώ σε διάφορα πράγματα που έχουν βραχυπρόθεσμη ισχύ. Υπάρχουν δράσεις οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν τάχιστα και θα μπορούσαν αυτές οι δράσεις α, να συνεχιστούν και στο μέλλον. Δεν εξαντλούνται βραχυπρόθεσμα μόνο. Παραδείγματο χάρη, για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την καταπολέμηση φτώχεια. Δεν είναι ότι δεν συμφωνώ. Απλώ θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διάφορες δράσεις, όχι μόνο μέσα στα πλαίσια ενός χρόνου, δηλαδή δεν πρέπει να εξαντλήσουμε και να ξεχάσουμε μετά, μετά από ένα χρόνο αυτό το θέμα, το θέμα της στόχιας δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνδεθεί από διάφορε, με διάφορες δράσεις στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα. Θέλω να πω στη συνάδελφό μου την κυρία Ντάνα. Το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Οι κοινωνικοί εταίροι, οι κυβερνήσεις, ε, τα πολιτικά κόμματα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Όταν μειώνεται ο πλούτος που παράγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, μπορεί να δημιουργήσει δυσκολία στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Και οι συντάξεις είναι ένα βασικό στοιχείο των δημοσίων πολιτικών σε οποιοδήποτε τμήμα του πλανήτη και πολύ περισσότερο στην γυραιά Ευρώπη, που έχει μια μακρά παράδοση προστασίας των πολιτών που παίρνει σάκα και οστά μέσα από το κράτος πρόνοιας, μέσα από το κράτος welfare. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που είπατε για τις, τους τρεις Εγώ όμως γιατί μίλησα για δύο πυλώνες, όχι γιατί διαφωνώ μαζί σας, αλλά γιατί. Πέρα από το δημόσιο πυλώνα, είναι λογικό και σωστό τα άτομα να έχουν και άλλες ευκαιρίες. Οικονομικής φύσεως, συμβατικής φύσεως. Και αυτή η διάκριση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πυλώνες σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν για λόγους καθαρά γλωσσικούς προσπάθησα να είμαι πιο συνοπτικός. το χάρη, κάποιος μπορεί να οικοδομήσει λίγο-λίγο τη σύνταξή του μέσω αποταμιεύσεων στην τράπεζα ή να έχει μία λύση συμβατική, συλλογική και κάθε φορά που, έχει, που υπάρχει μία μισθολογική αύξηση, ας πούμε, μπορεί ένα τμήμα αυτής της αύξησης, ας πούμε, να πηγαίνει στα συνταξιωτικά ταμεία για τη σύνταξή του. Επίσης, προσπάθησα να τονίσω και αν έχετε λύσεις να μου προτείνετε, είμαι στη διάθεσή σας για να βρούμε λύσεις. Πάντως, προσπάθησα να τονίσω το εξή. Η αναφορά στην φορολογική πολιτική για την προστασία των μισθών. Προφανώς υπάρχουν αυτόματοι τεχνικοί περιορισμοί. Παραδείγματο χάρη, για να εγγυηθούμε την αναπροσαρμογή των μισθών, θα πρέπει να υπάρχει προοδευτική φορολογική αύξηση. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κανένα συγκεκριμένο ε, μηχανισμό. Γιατί ουσιαστικά αυτοί οι μηχανισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εγώ μίλησα για την αρχή μονάχα. Καταλαβαίνω ότι όταν μιλάμε για τι αρχέ, <laughs> δημιουργούνται και αμφιβολίε. Ή για να μην πω υποψίε. Αλλά εγώ μίλησα για την αρχή και τίποτε άλλο. Ιδίω ό,τι αφορά την ε, αρχή τη ε, μισθολογική ισοτιμίας Ποια είναι αυτή η αρχή. Μπορούμε να ακούσουμε πολλές διαφορετικές γνώμες για είναι, αυτό, γιατί είναι αυτή η ισοτιμία. Και είναι πολύ λογικό να υπάρχουν διαφορετικές γνώμες. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε χώρα, λόγω της ιστορίας του, στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων, στις σχέσεις μεταξύ του κράτους και των ε, φορέων, των κοινωνικών φορέων, το θέμα της ισότητας ε, λύνεται με βάση την ε, συνείδηση που, έχει, που υπάρχει και, με βάση την πρακτική που υπάρχει. Επομένως, για λόγους πολιτικούς και πολιτιστικούς, υπάρχει μια συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα στην ε, εργασία και, στις, και στους μισθούς. Όπως και ανάμεσα στην ε, εργασία και στην παραγωγικότητα, που νομιμοποιεί την εργασία και την καθιστά αποτελεσματική. Γιατί σε ό,τι αφορά την ε, τροπολογία 19 για την παράγραφο 4, συμφωνώ, έχετε δίκο, δίκιο. Δείχνει με καλύτερο τρόπο αυτό που έγραψα εγώ ίδιος. Αν υπάρχει μια αμφισημία, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Πολύ Νομίζω ότι εντάξει, ε, ρεμισε Και ε, βασιζόμενοι εκεί θα ψηφίσουμε αύριο. Το σημείο 8 τώρα τη ημερήσιας διάταξης. Πασκάλ Γκρινί. Έχει το λόγο ο συνάδελφος για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση πρωτοβουλίας ε, για τα θέματα αυτά. Νέε μορφέ διαλόγου, άτυπε συμβάσει, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, ευελισφάλεια. Έχετε το λόγο. No. Σε σχέση με την ε, πρώτη σας παρουσίαση της έκθεσης πρωτοβουλίας σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή έρχεται σε μια χρονική περίοδο που ακολουθεί την κρίση, αλλά και προηγουμένως ήταν, πιστεύω, επίκαιρη αυτή η έκθεση, γιατί συμπίπτει με την αύξηση της ανεργίας και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε για τα θέματα αυτά της εξόδου από την κρίση, για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Υποδείγματος, ιδίως σε ό,τι αφορά την πλήρη απασχόληση, την βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να ευνοήσουμε μια πολιτική ποιοτική εργασία, την προσαρμογή της αγοράς εργασίας σε αυτούς τους στόχους και την ε, βελτίωση της δράσης μας κατά του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας στο βαθμό του δυνατού. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγές γραμμές, η δυνατότητα χρήσης των λεγόμενων ατυπικών συμβάσεων που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και αυτό οφείλεται πιστεύω στην κρίση, την οικονομική που διερχόμαστε, είναι απαραίτητο εδώ να θέσουμε επιτάπητος τα υπέρ και τα κατά αυτών των συμβάσεων, αυτά από τα οποία αναμένουμε <clears throat> από τις θέσεις αυτές εργασίες και επίσης σε σχέση με την δυνατότητα προστασίας των εργαζομένων που βρίσκονται σε τέτοιου είδους ατυπικές Σχέσει εργασία και να ζητήσουμε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να εξετάσουν το θέμα αυτό και να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει και η σωστή εφαρμογή των συμπεφωνημένων σε ό,τι αφορά την ευέλικτη ασφάλεια. Ο κύριο στόχο αυτή τη εκθέση πρωτοβουλία ούτω ή άλλω είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον διεισμό τη αγορά εργασία, μεταξύ μια σταθερή δύναμη εργασία και τη λεγόμενη εφήμερη εργασία, που είναι η επισφαλής αυτές ε, θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι πολύ πιο ευέλικτες. Στην έκθεσή μου λοιπόν, εγώ προσπάθησα να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα σε τρία αλληλένδετα τμήματα, καταρχήν τις ατυπικές συμβάσεις, για τις οποίες πιστεύω να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στα διάφορα κράτη-μέλη, στην περίπτωση της Δανίας, θα πρέπει να ενισχύσουμε <clears throat> την προστασία των εργαζομένων μέσα σε αυτό το πιο εύκαμπτο πλαίσιο αλλά με ενεργές πολιτικές αγοράς εργασίας θα πρέπει επίσης να κάνουμε μια προσπάθεια να συνενώσουμε τις διάφορες μορφές των ατυπικών συμβάσεων γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίε αυτού του είδους. Επίσης <clears throat> θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι μπορεί να είναι απαραίτητες αυτές οι ατυπικές συμβάσεις για άτομα τα οποία είναι άνεργα, γιατί θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτούς οι οποίοι χάνουν τη θέση εργασία τους να επανέλθουν το ταχύτερο δυνατό σε μια θέση απασχόλησης. Οι στατιστικές καταδεικνύουν ότι όσο πιο μεγάλο χρόνο μένει κανείς έξω από την αγορά της εργασίας, τόσο πιο δύσκολο είναι να επανέλθει σε μια θέση απασχόλησης ακόμα και με ατυπική σύμβαση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διατηρήσει κανείς κάποια παρουσία στο χώρο εργασίας, ακόμα και ατυπικού χαρακτήρα. Επίσης, οι ατυπικές συμβάσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την παράνομη η μαύρη εργασία που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο τμήμα ειναι η αντιμετώπιση της ευέλικης ασφάλειας και το θέμα της εξασφαλισμένης επαγγελματικής καριέρας εδώ πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι επιχειρήσεις όταν δεν έχουν πολλές οικονομικές προοπτικές και αυτό είναι ακόμα χειρότερο σήμερα από τις άλλες εποχές, όταν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης λοιπόν σε σχέση με το μέλλον, προτιμούν να μην προσλάβουν άτομα με σταθερές σχέσεις εργασίας, να τους αρνηθούν λοιπόν την πρόσληψη, γιατί φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν στο μέλλον να διατηρήσουν τη δύναμη εργασίας τους. Αυτό επομένως είναι κάτι το αρνητικό. Θα πρέπει αντίθετα να προωθήσουμε την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή να μπορέσουν εκεί οι επιχειρήσεις να έχουν εμπιστοσύνη και οι άνεργοι να μπορέσουν να ξαναβρούν θέσεις εργασίας. Η έννοια λοιπόν αυτή της ευέλικης ασφάλειας μπορεί να δώσει μια στιγμιαία απάντηση σε αυτό το άγχος που νιώθουν οι επιχειρήσεις ενώπιον της κρίσης. Αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε στο μυαλό μας ότι οι συμβάσεις αορίστου χρόνου θα πρέπει να είναι ο κύριος κανόνας, θα πρέπει να είναι η φυσιολογική κατάσταση στο, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις εργασίας, εκτός αν ο εργαζόμενος θέλει να προχωρήσει σε κάποια μορφή κατάρτισης ή αν θέλει να αποχωρήσει για λόγους οικογενειακούς, προσωρινά κτλ. Θα πρέπει επομένως να καταδικάσουμε την καταχρηστική αντικατάσταση των σταθερών σχέσεων εργασίας με ατυπικές συμβάσεις. Αυτό λοιπόν είναι μία από τις βασικές δυσκολίες που έχουμε να κάνουμε τις ατυπικές συμβάσεις και θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των ατόμων που εργάζονται με ατυπικές μορφές συμβάσεων με την απαραίτητη προστασία σε κοινωνικό επίπεδο προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Τρίτο τμήμα τη έκθεση είναι ο κοινωνικό διάλογο. Είναι απαράγραπτος ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων εδώ, στα κράτη-μέλη μας. Δεν είμαστε πάντα στο επίπεδο κοινωνικού διαλόγου. Πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν και ο κοινωνικός διάλογος για την απαραίτητο και το βλέπουμε όλο και περισσότερο για τέτοιες μορφές συμβάσεων, αλλά εξάλλου αυτό εφαρμόζεται και στο σύνολο όλων των σχέσεων εργασίας που μπορούν να υφίστανται στα κράτη-μέλη μας και στην προβληματική της ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί λοιπόν ο κοινωνικός διάλογος <clears throat> και να επεκταθεί στο σύνολο των κρατών μελών. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Θα προχωρήσουμε με ένα καινούριο τρόπο. πίσω από αυτή την εκθεσή σας. Θα θυμάστε την πρώτη μελέτη εδώ σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου, την ίδια που είχατε παρουσιάσει στο τέλος της προηγούμενης θητείας του Κοινοβουλίου. Αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν ένα συνδετικό κρίκο για παροτριντικά στοιχεία για το σύνολο της εργασίας μας. Και βάσει της μελέτης αυτής ε, θελήσαμε ακριβώ να αναλάβουμε αυτή, να συντάξουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι το εξετάσατε το υλικό σχετικό και οι συνάδελφοι επίσης αναφέρονται σε αυτά. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία σε αυτά. Για να δούμε τώρα για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να μας ακούσουν εδώ από την Επιτροπή μας βάσει των δύο μελετών που έχουν συνταχθεί και πριν να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο μάλλον στην εργασία της όλης επεξεργασίας ε, για την ε, πρόταση της κ. Γκρανή. Η εκπρόσωπος ε, η κυρία Ελίζαμπεθ Μπιλέτα έχει το λόγο για να μας μιλήσει, να μας παρουσιάσει τις δύο μελέτες που έχουν συντάξει και τα κύρια στοιχεία δε των μελετών αυτών σας έχουν ήδη δοθεί. Η κυρία Μπιλέτα έχει το λόγο λοιπόν, δέκα λεπτά μόνο και οι δύο μελέτες έχουν σαν θέμα το ένα flexible form of work κλπ. Σχετικά με την ατυπική εργασία και το άλλο exploratory analysis κλπ σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, μελέτη κλπ. Έχετε το λόγο κυρία μου για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ Σας ευχαριστώ για την ε, θετική υποδοχή που δίνετε στην έρευνά μας. Θα ήθελα απλώς να, να παρουσιάσω καταρχήν τα όρια αυτής της έρευνας. Εμείς εστιάσαμε την προσοχή μας σε πολύ ατυπικές μορφές εργασίας και προσπαθήσαμε να ατενίσουμε αυτή τη μορφή αυτό το ειδικό τμήμα της αγοράς εργασίας. Και σας ε, τονίζω ότι εδώ μας ενδιαφέρουν πολύ βραχυπρόθεσμες θέσεις εργασίας που έχουν διάρκεια λιγότερο από έξι ε, μήνες μερική εργασία λιγότερο των 10 ωρών και σχέσεις οι οποίες είναι ουσιαστικά σχέσεις εφημερίας και όχι σταθερής εργασίας. Είναι ατυπικές σχέσεις εργασίας, δεν πειράζει παρόλα αυτά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτό το οποίο θέλω να πω, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε τέτοιου είδους σχέσεις εργασίας όταν ακόμα οι περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται στις κανονικές σχέσεις εργασίας. Σε μία από τις μελέτες μας είδαμε ότι 76% των εργαζομένων είναι ακόμα σε παραδοσιακές, μακρού χαρακτήρα, μόνιμες σχέσεις εργασίας. Γιατί ατενίζει αυτό το τμήμα συμβάσεων βραχαίως χρόνου. Πολλοί λόγοι υπάρχουν. Ένας από αυτούς τους λόγους, και το είπε η κυρία εισηγήτρια προηγουμένως, ο λόγος είναι ότι η τάση είναι προς την αύξηση των μορφών εργασίας βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Υπάρχει μια σημαντική αύξηση και επομένως χρήζει περαιτέρω εποπτεία σε αυτό το τμήμα. Άλλος λόγος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά αυτός ο σεβασμός είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη για τουλάχιστον τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος, και το έχουμε δει ήδη, είναι ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιου είδους πολύ συγκεκριμένων συμβατικών εργασιακών σχέσεων. Υπάρχει λοιπόν ένας σημαντικός ρόλος τον οποίο θα πρέπει να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι όταν πρόκειται για συγκεκριμένες μόρφες προσωρινής εργασίας ή σταθερής εργασίας που έχουν πολύ βραχή χρόνο και που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Μια δεύτερη πτυχή, ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο αυτές οι πολύ πολύ ατυπικές συμβατικές σχέσεις παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι ότι η αντιπροσωπευτικότητα και η αντιπροσώπευση αυτών των εργαζομένων σε επίπεδο συνδικαλιστικό δεν έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα λόγω του προφίλ που παρουσιάσουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς λόγω της ε, γεωγραφικής ε, τοποθέτησης του χώρου εργασίας. Δεν έχει αναπτυχθεί διότι πολλές φορές δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των ατυπικών εργαζομένων. Υπάρχει λοιπόν πολλή χώρο για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την ενίσχυση τη ικανότητα των κοινωνικών εταίρων και θα σα είπα ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μονάχα στα κράτη-μέλη, <clears throat> τα οποία εισήλθανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από το 2004, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια ανησυχητικά μηνύματα σε χώρες όπως και η Δανημαρκία, όπου τα εργασιακά συνδικάτα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση της σύνολης εργατικής δύναμης και υπάρχει μείωση του αριθμού των μελών τους που θα μπορούσαν να υποσκάψουν την νομιμοποίηση των εργατικών ενώσεων ω κοινωνικών εταίρων μέσα στα πλαίσια τη συζήτηση για την ευελίξη ασφάλεια, ακόμα και στην Δανία. Βέβαια, παράλληλα, υπάρχει ελάχιστα ανεπτυγμένος έλεγχος της εφαρμογής των δικαιωμάτων των εργαζομένων για αυτούς τους ατυπικούς εργαζομένους, λόγω της έλλειψης ικανότητας της επιθεώρησης εργασίας σε πολλά από τα κράτη-μέλη. Γιατί όμως και πάλι να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το μικρό, το κούτσικο τμήμα του εργασιακού πληθυσμού. Αυτό γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ένδυας, ένδυας ενώ εργάζονται, η ένδυα των εργαζομένων. Αυτό είναι μια ειδική πτυχή, αν εξετάσουμε το εισόδημα των οικοκυριών αυτών των εργαζομένων. Δεν είναι τόσο οι άμεσες αποδοχές αυτών των εργαζομένων ακόμα και σε αυτές τις ο, πόσο ατυπικές μορφές εργασίας που υπόκεινται σε κινδύνους και σε απειλές. Όχι, είναι περισσότερο το μακροπρόθεσμο, το προοπτικό θέμα, το γεγονός ότι αυτές οι τόσο ατυπικές ρυθμίσεις εργασίας δεν θα ειδύναντο να οικοδομήσουν δικαιώματα συνταξιοδοτικά, δικαιώματα για επιδόματα ανεργίας, δικαιώματα για υγειονομική υπερίθαλψη. Ένα μείζον πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό για τα λεγόμενα ε, συστήματα mini-jobs στην Γερμανία, όπου δεν υποχρεωτική η ασφάλιση των εργαζομένων και όπου οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι θα πρέπει να αυτοασφαλιστούν ιδιωτικά. Και αυτή η ιδιωτική ασφάλιση Επίσης είναι ένα υψηλό κόστος. Και εξάλλου δεν είναι ο κίνδυνος αυτός κάθε αυτός σε ό,τι αφορά αυτές τις ατυπικές μορφές εργασίας. Ίσως είναι περισσότερο εκτεθειμένοι αυτοί οι εργαζόμενοι από αυτούς που έχουν μια μόνιμη σχέση εργασίας. Όχι, είναι ο συνδυασμός μιας αυξημένης έκθεσης στον κίνδυνο και της μείωσης της κοινωνικής κάλυψης που κάνει αυτού του είδους τις συμβατικές σχέσεις να είναι μακροπρόθεσμα ιδιαίτερα επισφαλείς και επικίνδυνες και όπου πολλές φορές βλέπουμε εκ των υστέρων τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μετά και τη λήξη της σύμβασης για τις ρυθμίσεις ευέλικης ασφάλειας. Θέλω να το δύο σημεία. Τι είναι η ασφάλεια αφενός, τι είναι η ευελιξία από την άλλη πλευρά. Αυτό το οποίο έχουμε δει μέσα από πολλές από τις μελέτες μας είναι ότι η ασφάλεια ή η ανασφάλεια είναι κάτι το οποίο σωρεύεται. Έχει κανείς χαμηλά προσόντα, χαμηλές δεξιότητες, εργάζεται σε δουλειές χαμηλής εξειδίκευσης με χαμηλές αποδοχές. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία αυξάνουν την ανασφάλεια στο χώρο εργασίας. Αλλά δεν εξετάζει κανείς στο ίδιο επίπεδο την ασφάλεια και την ανασφάλεια. Αν δούμε μια πορτογαλική μελέτη η οποία έλαβε χώρα σε σχέση με το συγκεκριμένο ερώτημα του αν ένας εργαζόμενος νιώθει ασφαλής στην εργασία του. Και προφανώς κάποιος ο οποίος έχει μια μόνιμη σχέση εργασίας νιώθει ασφαλέστερος από αυτούς οι οποίοι εργάζονται λιγότερο από 34 ώρες την εβδομάδα. Μόλον τούτο υπήρχαν εργαζόμενοι οι οποίοι δούλευαν λιγότερο από 15 ώρες την εβδομάδα οι οποίοι ένιωθαν πάρα πολύ αρκετά ασφαλείς. Και εδώ θα η τι να πει ότι κάποιοι από αυτούς τους εργαζόμενους επιλέγουν αυτή τη μορφή σχέσεως εργασίας ατυπικού χαρακτήρα συμβατικού δε. Παρόλα αυτά, τέτοιου είδους επιλογές θα πρέπει να εξεταστούν πάρα πολύ προσεκτικά, ιδίω όταν βλέπουμε τι μπορεί να επιλέξουν μέσα εισαγωγικά οι γυναίκες προσπαθών να συνδυάσουν τον οικογενειακό χώρο με τον χώρο εργασίας. Τέτοιου είδους ασφάλεια λοιπόν είναι σχετικού χαρακτήρος, όχι σχετικού χαρακτήρα και μόνο επειδή υπάρχει ετερογένεια στις συμβατικές σχέσεις των εργαζομένων αυτών, αλλά σχετική ακόμα και λόγω του κοινωνικού περίγυρου. Και στις κάτω χώρες δεν θεωρεί ότι, ο κόσμος δεν θεωρεί ότι το να είναι κανείς σε μια τέτοια ατυπική σχέση εργασίας είναι επισφαλές, όπως σε άλλες χώρες ή σε άλλες κοινωνίες. Και πάλι, τι είναι η ασφάλεια. Συγγνώμη, τι είναι η ευελιξία οι οργανώσει των των εργαζομένων πολλές φορές μπορούν να γελιογραφηθούν των εργοδοτών, συγγνώμη. Γιατί μπορεί να θεωρηθούν ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι η ευελιξία και μόνο η ευελιξία. Ενώ η μελέτη μας έδειξε ότι υπήρχαν κάποιες οργανώσεις εργοδοτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι θεωρούσαν ότι ενδεχομένω υπάρχουν κάποια όρια προς το συμφέρον της ίδιας της επιχείρησης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ευελιξίας ασφάλειας. Το είδαμε αυτό στο ακριτικό Λουξεμβούργο, στην Ουγγαρία και στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου οι εργοδότες αντιδρούσαν στην υπερβολική ευελιξία ασφάλεια και θεώρησαν ότι η άμετρη αύξηση της εργασίας με μερική απασχόληση και των επισφαλών μη συμβατικών σχέσεων εργασίας θα είναι δύνατο να έχει και ένα αρνητικό αντίκτυπο και δυσβάστακτο κόστος για την επιχείρησή τους, η οποία θα καθίστατο μη αποδοτική και αποτελεσματική και θα εμείωνε την απόδοση αυτή τη επιχείρηση. Μήπω μπορώ να σα ζητήσω να κλείνετε, λέει η πρόεδρο, να τελειώσετε κάποια στιγμή. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Κλείνον, θα ήθελα να τονίσω ότι ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες πολιτικές που χρειάζονται και οι οποίες συνδέονται με πολιτικές πρόληψης και που συνδέονται με πολιτικές εκπαιδευτικού χαρακτήρα για να μειώσουν την σχολική αποτυχία και τα άτομα με χαμηλά προσόντα, και για την πρόληψη του κινδύνου απώλειας εργασίας, θα πρέπει οι πολιτικές ευελιξίας να βασίζονται στο μακροπρόθεσμο και στο επέκεινα και να δουν τι γίνεται μετά από τη σύναψη μιας συμβατικής σχέσης για τους εργαζόμενους και στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξουν συντετονισμένες πολιτικές μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν το τοπικό επίπεδο και να οικοδομούν σε τοπικό επίπεδο απαντήσεις για τους εργαζόμενους που ίσως και πάλι μπορεί να αποτελούν σήμερα ένα πολύ μικρό τμήμα της αγοράς εργασίας, αλλά όλο και περισσότερο αυξάνονται και πληθύνονται. Ευχαριστώ. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της ανταλλαγής απόψεων. Μετά την παρουσίαση της συζητήτριας. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στο Business Europe ε, που εκπροσωπεί τους κοινωνικούς εταίρους, Μαξίμ Σερούτη, ε, ε, σύμβουλος για τέτοια θέματα, για κοινωνικά θέματα. κυρία Πρόεδρε, Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μας αρέσει ο διάλογος με την Επιτροπή σας και θα ήθελα να το πω αυτό πριν ξεκινήσω την παρέμβασή μου. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια τα οποία συνδέονται με το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Γκρουνή που λάβαμε πριν τη συνεδρίαση αυτή και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι νομίζω πως ο τρόπος με τον οποίο είναι συνταγμένη η έκθεση είναι πολύ ισορροπημένος και αντανακλά τις διαφορετικές ε, καταστάσεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι καλό σημείο αφετηρίας λοιπόν. Μας αρέσει το γεγονός ότι εστιάζει η έκθεση στην ανάγκη να δημιουργηθεί, να τονωθούν οι θέσεις απασχόλησης, να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Και αναφέρεται επίσης στην ε, συζήτηση που γίνεται για την στρατηγική Ευρώπη 2020 και για τους υπολογισμούς που γίνονται ε, και τις ε, συνέπειες από τη μεγαλύτερη δημιουργία θέση απασχόλησης. Παραδείγματο χάρη, αν από 1% πάμε σε 2% ρυθμό ανα, οικονομικής ανάπτυξης, θα δημιουργηθούν 6,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Η έκθεση τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και τα μέτρα που σκοπό έχουν να μειωθεί το διοικητικό άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά να απλουστευθούν ε, οι διατυπώσεις ε, για την πρώτη πρόσληψη. Αυτό είναι καλό που υπάρχει στην έκθεση. Μου αρέσει επίσης η έμφαση που δίνεται στην ευέλικτη ασφάλεια και στην ανάγκη τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, κάποιες πασαρέλες εύελιξης ασφάλειας. Μ' αρέσει επίσης το γεγονός ότι η έκθεση δείχνει ότι η ευελιξιασφάλεια είναι σημαντική όταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι καλή και όταν υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχει ψηλότερη ανάγκη ευελιξης ασφάλειας, λόγω ακριβώς των δυσκολιών. Και νομίζω ότι αυτό έδειξε η κρίση στην Ευρώπη. Η... Τα συνδικάτα των εργαζομένων με των εργοδοτών σε συζητήσεις που έκαναν ε, κατάφεραν να μειώσουν ε, τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που χάνονται. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν τέτοια μέτρα διαλόγου εργοδοτών εργαζομένων. Ε, σημαντικό στοιχείο των εθνικών μεταρρυθμίσεων θα είναι να βοηθήσουν τους εργαζόμενους για να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς. Επίσης, ένας πολύ σημαντικό ρόλος ε, θα μπορούσε να δοθεί στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση με μεγαλύτερες επενδύσεις ε, σε αυτές. Ε, θα ήθελα να τονίσω την έκθεση του Eurofound της περσινής χρονιάς που λέει ότι τα τρία των επιχειρήσεων έχουν ήδη ένα συστηματικό τρόπο για να συμπεριλάβουν την κατάρτιση στις δραστηριότητε τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Ε, δηλαδή οι επιχειρήσεις ε, παίρνουν την κατάρτιση πραγματικά στα σοβαρά. Και εμείς θα πρέπει να τονίσουμε την ε, ανάγκη τα άτομα να κινητοποιηθούν για να μαθαίνουν προκειμένου να κρατήσουν τη δουλειά τους. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό πέρα από τις δράσεις, τις όποιες δράσεις προωθήσουν οι επιχειρήσεις. Επίσης, θα ήθελα να αντιδράσω στην έκθεση, εκεί που λέει ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Προφανώς θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και, εργαζομένων ε, μπορούν να προωθήσουν καλές λύσεις και να βελτιώσουν την κατάσταση στην ε, αγορά εργασίας. Πρόσφατα ε, τελειώσαμε τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες πλαίσιο για την αγορά εργασίας που ελπίζουμε ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στα κράτη-μέλη και θα βοηθήσει τη συζήτηση για τις εθνικές μεταρρυθμίσεις. Φυσικά ένα στοιχείο είναι ότι θα παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση στην ε, τριμερή Σύνοδο Κορυφής 25 Μαρτίου. Νομίζω ότι είναι ένα επίτευγμα των, των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και δείχνει πόσο πραγματικά θέλουμε να συνεισφέρουμε στην όλη προσπάθεια. Θα ήθελα να κάνω τώρα και άλλα σχόλια που συνδέονται με την ε, ασφάλεια στην αγορά εργασία Και τι είναι αυτή η ασφάλεια. Η προηγούμενη ομιλήτρια είπε διάφορα πράγματα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η ικανότητα των ατόμων να διατηρήσουν ή να ενδυναμώσουν την απασχολησιμότητά τους και να δράξουν νέες ε, ευκαιρίες απασχολησιμότητας στη δουλειά, ε, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Μαζί με τις ευκαιρίες για κατάρτιση, στις οποίες αναφέρθηκα, ε, όλα αυτά έχουν σαν σκοπό να προωθήσουν την κινητικότητα στην αγορά εργασίας της Ευρώπης. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχει και, υπάρχουν και ευέλικτα συμβόλαια εργασίας. Η έκθεση μιλάει για αυτά, τα ευέλικτα συμβόλαια και με το χαρακτηρισμό όμως ε, των συμβολέων αυτών, των συμβάσεων αυτών ως ε, ατυπικών, αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό που είπε η κυρία Μπιλέτα. Μας είπε η κυρία Μπιλέτα ότι 76% των συμβάσεων εργασία είναι τυπικές συμβάσεις. Εγώ νομίζω ότι είναι χαμηλότερο το ποσοστό, γύρω στο 50% κινείται. Ε, νομίζω ότι οι ατυπικές μορφές εργασίας έχουν αυξηθεί. Ε, δεν είναι κάτι περιορισμένο λοιπόν. Δύο καταληκτικές παρατηρήσεις. Ε, για τους νέους στην αγορά εργασίας. Νομίζω είναι προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε Ε, την, ε, τους νέους ε, στην εργασία. πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτούς που φεύγουν νωρίς από το σχολείο. Ένα στους 7 φεύγει νωρίς, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για τις ευέλικτες μορφές εργασίας θέλω να τονίσω ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε, αυτές οι μορφές εργασίας ανταποκρίνονται και στις προτιμήσεις των ατόμων και στο μεγάλο βαθμό ατομικότητας που υπάρχει. Ε, το 80% των εργαζομένων που είχαν ερωτηθεί το 2005 είχαν πει ότι ήταν ικανοποιημένοι το, με τις συνθήκες εργασίας τους. Και το 76% που δουλεύουν με μερικό χρόνο απασχόλησης επιλέγουν να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Το πιο σημαντικό καταληκτικά είναι να κλείσουμε το χάσμα μεταξύ των ευέλικτων μορφών εργασίας και των μόνιμων μορφών απασχόλησης. Γιατί αυτός ο κατακαιρματισμό στην αγορά εργασίας είναι μεγάλο πρόσκομα στη δημιουργία απασχόλησης, θέσεων απασχόλησης. Ε, στις χώρες όπου, όπως στην Ολλανδία ή στη Δανία, αυτές τις ατυπικές μορφές απασχόλησης τις βλέπουν θετικά, εκεί ακριβώς οι άνθρωποι που δουλεύουν με διαφορετικού είδου τελικά έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ε, αυτά και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κ. Τζόντε Καϊόν έχει το λόγο. Πέντε λεπτά έχετε στη διάθεσή σας και καταλάβατε ότι η συγγήτριά μας ε, παρουσίασε σε τρία μέρη αυτό ε, για τις άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, ε, ασφάλεια και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου και θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας καλέσατε για να εκφράσουμε την απόψή μας. Εδώ να σας πω ότι πολλά ερωτηματικά είχαμε για την έκθεση αυτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τι θα βοηθήσει τι θα χρησιμεύσει για τη ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι κάπως ασαφές. Υπάρχουν τρομερές φιλοδοξίες που έχουμε την ευελασφάλεια, τις άτυπες συμβάσεις. Το δεύτερο αυτό το ευελασφάλεια είναι πολύ, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο αλλά και απλό ένα μέρος της συζήτησης, πνιγενική συζήτηση, μας βάζει μετά σε ειδική συζήτηση και εκεί γίνεται τρομερή η δυσκολία. Για να δούμε τώρα μετά από όλα αυτά. Κάτι το προκατερτικό. Η ευελίξη ασφάλεια είναι κάτι που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα με την κρίση, έχει να κάνει με πάρα πολλά εκατομμύρια κόσμο τώρα που έχουν προβλήματα ε, 30% σε μερικές χώρες είναι εδώ που έχουν πρόβλημα εργασίας. Και όπως είπαμε προηγουμένως εδώ έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο και έφραυστο χαρακτήρα. Γι' αυτό ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να απαντήσει σε όλα αυτά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καλέσει τις διάφορες χώρες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, να έχουν υποχρεώσεις και ένα μέρος εδώ από την έκθεση ακριβώς έχει να κάνει με αυτό. Είτε Ανακατεύοντα την ασφάλεια και τις άτυπες συμβάσει, ε, ιδιαίτερα δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ποιο είναι όλος στόχος όλων αυτών των εργειών για τις ε, άτυπες ε, συμβάσει. Εντάξει, δεν θα σα κάνω να κλάψετε, είναι άσκημη κατάσταση. Εδώ η Σομπνάκ κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που είπε ότι θέλησε να βουτήξει σε αυτόν τον κόσμο και μόλις ε, ε, θα βρω ένα ε, κατάλληλο συμβόλαιο που να μιλάει για δυόμιση ώρες δουλειά άτυπη εργασία, σύμβαση εργασίας, τότε θα σταματήσω να ψάχνω. Και το βρήκε αυτό. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε αυτή τη μορφή εργασίας θα τη δεχτούμε είτε θα δούμε διάφορες άλλες μορφές κοινωνικής συνεργασίας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά χρειάζονται και μία ανάλυση, βάθηση πάνω σε διάφορες πτυχές. Θα δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Κάτι ακόμα στην ευελίξη ασφάλεια. Εδώ είχαμε και μια συζήτηση με την έκθεση που έγινε από το Ίδρυμα του Δουβλίνου. Είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε σε συγκεκριμένα σαφή πράγματα σχετικά με την ευελίξη ασφαλεία. Πρώτη ευθύνη ακριβώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εφαρμοστεί το κοινωνικό δίκαιο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πρώτη ευθύνη επίσης και υποχρέωση και του Ευρωκοινοβουλίου, των συνδικάτων, των κοινωνικών εταίρων. Έτσι επίπεδο, γιατί είναι τρομερό πρόβλημα ο παράνομα εργαζόμενος ε, και το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε αυτά το σύστημα για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μορφή εργασία και επίση στι οικοδομέ. Ξεκίνησε μια εκστρατεία σχετικά εκεί. Υπάρχει μια, υπάρχουν αντιμετωπίσει όταν λοιπόν, έχουμε παράνομη εργασία, περισσότερο αντιπίσυβαση δεν είναι ανακάτεμα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των ταμείων, των διαχωτικών κλπ. στην πολιτική που θέλει να ασκήσει θα πρέπει να προσπαθήσει ώστε να ισχύσει το δίκαιο. Σε ορισμένα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το 40% του ΑΕΠ που, είναι, που έχει να κάνει με την παράνομη εργασία. Και έχουμε μια ευελιξία του χρόνου εργασία, διαπραγματευόμαστε και χρόνια και σχετικά με τις αμοιβέ. Το νόημα είναι υπαρξιακό τη ε, από το 17ο αιώνα. Δεν το ανακαλύψαμε σήμερα. Είχαμε, ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ε, για τον χρόνο εργασία κλπ. κλπ. Δεν σα λέω λεπτομέρειε. Έχουμε λοιπόν αυτή την εσωτερική ασφάλεια το έχουμε πει, το έχει πει και ο εκπρόσωπο από το Ίδρυμα του Δουβλίνου, για αυτή την εσωτερική και για την μερική ανεργία όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν ισχύουν παράμετροι οι οποίε μπορούν να προσφέρουν ορισμένε εγγυώσει. για να το πρόβλημα και τι γίνεται, πού είναι πρόβλημα η ευλεξασφαλιακή Δανία ακόμα γιατί με τις Δανού συζήτησα χθε ότι εδώ από με μεταβατική περίοδο ε, αυτή είναι ιδιαίτερα μακρά σε μια παρόμοια κρίση και στη συζήτηση που γίνεται στη Γαλλία, διακρίνεται Γαλλία τι είναι, Πώ θα προστατευθούν οι άνεργοι γιατί δεν θα έχουν πια ε, επιδόματα. Τι γίνεται, όλα αυτά, η όλη διαχείριση και αυτά είναι στην κοινή μα έκθεση. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρω σήμερα βρίσκονται στην έκθεση αυτή για του από του κοινικού εταίρου αυτή. Η κοινή του εγγύηση που λέει ότι θα πρέπει να τα εξασφαλίσουμε όλα αυτά. Θα κατάλληλα αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε κατάλληλο τρόπο αυτή τη μεταβατική περίοδο, η οποία είναι, η οποία είναι πολύ μπερδεμένη για τη διαχείρισή τη, γιατί πολλά κοστίζει. Για να δούμε λοιπόν. Αυτή η ευελιξασφάλεια σε αυτή τη μεταβατική περίοδο θέλει μια επιβολή φόρου και μια αναδιανομή και αυτό είναι σημαντικό μέρος. Εάν παραστήσουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, εντάξει, ρεμούμε, η κοινωνική εταιρεία φταίνει, ναι, αλλά τι κάνουν μετά αυτοί, τι θα κάνουν αυτοί στη μεταβατική περίοδο, ποια είναι τα μέσα τώρα για να μπορέσουμε ε, αυτή και την κατάρτιση να εξασφαλίσουμε και τη μεταβατική περίοδο. Για να δούμε στι πραγματεύσει στην κάθε χώρα, να δούμε όμω και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προσκαλέσουμε αυτών των ταμείων μια αλλαγή σε σχέση με αυτή τη μεταβατική περίοδο. Τώρα στη συζήτηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο αν θέλουμε να είναι κάτι το δυνατό για να βοηθούν τα κράτη να λύσουν τα προβλήματά τους εκεί που υπάρχουν διαφορές στις κοινωνικές σχέσεις, εντάξει τα συμμερίζουμε όλα αυτά και ο κοινωνικός διάλογος στις ορισμένες χώρες είναι, δεν υπάρχει καθόλου σήμερα. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να βρούμε και τους ε, συνδικαλιστές και τους εργοδότες των Ατάλλων. Χρειάζεται αυτά τα μέσα, τα εργαλεία να ενισχυθούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να παροτρύνει τους πολιτικούς να τα κάνουν αυτά πραγματικότητα. Εάν ε, παραμένουμε έτσι σε αυτό το γενική έννοια της ασφάλεια ω είναι κείμενο βλέπω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ένα κείμενο που να μην υπάρχει αυτή η λέξη. Είναι χαρακτηριστικό σύμβολο τη Ευρώπη. πια αυτό το ασφάλεια Είναι σύμβολο αναγνώριση ποιοτικού προϊόντο. Δεν ξέρω αν είναι ποιοτικό αυτό προϊόν, τέλο πάντων. Ε, ε, πρόκειται για σημείο αναφορά. Αλλά σα παρακαλώ προσπαθήσουμε να εργαστούμε. Εμεί προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Και βλέποντα σε αυτό το κοινοκείμενο των κοινωνικών εταίρων ε, είναι αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ασχολούνται όλοι με αυτό και θέλουμε να του βάλουμε κάθε σάλτσα σε κάθε περίπτωση. Ε, θα προκύψει μία απόρριψη, να το καταλάβουμε αυτό. Και θα γίνει αυτό. Προσπαθεί κανεί να δικαιωθεί τα δικαιολόγητα μέσα τη χρησιμοποίηση τη αφελού αυτή τη έννοια. Ε, και αντί να έχουμε μια σωστή συζήτηση πλούσια, θα έχουμε μια φτωχή συζήτηση σας ευχαριστώ για να σας έχω πληροφορημένους. Θα ήθελα να αναφέρω στα μέλη της ε, Επιτροπής μας ότι έχουμε συμφωνήσει για την αρχή αυτής της έκθεσης. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας και επομένως έχετε κάθε δικαίωμα να ρωτάτε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της έκθεσης και ποιο θα είναι το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης μέσα στο Κοινοβούλιο μας για αυτή την έκθεση, η οποία είναι σημαντική για μας και θέλουμε να υπάρξει μια συλλογική συζήτηση όπου να παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο και η Επιτροπή μας, δηλαδή να είναι μια έκθεση πρωτοβουλία η οποία θα επιτρέψει επί τη βάση των συμπερασμάτων της που θα εγκριθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παροτρύνει την Κομισιόν να προχωρήσει στις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Για το συγκεκριμένο σημείο της ευέλιξης ασφάλειας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο λόγος ύπαρξης ουσιαστικά αυτής της έκθεσης είναι η συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στη μελέτη η οποία μας παρουσιάστηκε για τον αντίκτυπο νέων μορφών εργασιακών σχέσεων και για την εξέλιξη του εργασιακού δικαίου στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συντάχθηκε από την Ένωση για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Εργασίας και την Ένωση για τις Εργασιακές Σχέσεις και η αρχή, στην αρχή δεν υπήρχε καθόλου η έννοια της ευελίξης ασφάλειας μέσα σε αυτή την έκθεση, μονάχα μετά από τη διαπραγμάτευση των πολιτικών ομάδων παρισέφρισε αυτή η διατύπωση, ακόμα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής συζήτησης ακόμα και τώρα. Λοιπόν, ανοίγω τη συζήτηση μετά από όλα αυτά. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Τόμας Χέντελ. Εγώ μπορώ να αποδεχθώ πολλά από αυτά τα οποία ανέφερε η συγγήτρια. Ε, αλλά όχι όλα, γιατί αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να πάρω το λόγο. Πέντε παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την εισηγήτρια ότι σε ό,τι αφορά μια στρατηγική απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να περιοριστούμε μονάχα σε θέσεις ποιότητος, αλλά θα πρέπει να είναι θέσεις σταθερές και μόνιμες. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την εισηγήτρια να αναφέρει αυτό το σημείο, να υπάρξει απαραίτητη προσθήκη στο σημείο 13, ώστε να διατυπωθεί και πάλι το αίτημά μας να υπάρχουν σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας. Δεύτερη παρατήρηση. Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό της ευελιξασφάλειας και της στρατηγικής απασχόλησης δεν αναφέρεται στην έκθεση το γεγονός ότι αυτή η στρατηγική τα τελευταία χρόνια οδήγησε στο να είναι οι ατυπικέ και επισφαλείς θέσει εργασία ένα τομέα ο οποίος αυξήθηκε κατά 60%. Αυτό δεν είναι δάφνες τις οποίες έδρεψε η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης, γιατί αυτή η πολιτική συνδέεται με υπερβολική ευελιξία και ελάχιστη ασφάλεια. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν στο σημείο 14 να υπάρξει μια διατύπωση, μια πρόσθετη διατύπωση που θα αναφέρει αυτό το στοιχείο. Στη συνέχεια, στο σημείο 15, γίνεται σαφές ότι η ευελιξασφάλεια δεν προέρχεται από μια συνένεση των κοινωνικών εταίρων, αλλά Αντίθετα, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια καλύτερη εξασφάλιση σε κοινωνικό επίπεδο των εργαζομένων που υπόκεινται σε αυτή τη μορφή εργασίας. Τέταρτη παρατήρηση. Θεωρώ θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να σκεφτούμε καλύτερα για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με ατυπικές μορφές εργασίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδικαιολόγητο αυτό το οποίο λέγεται στο 29 για τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτή την περίπτωση ότι και η Κομισιόν και οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να προσκληθούν και να παροτρινθούν να βελτιώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ατυπικές μορφές εργασίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν συμβάσεις οι οποίες οδηγούν σε κοινωνικό ντάμπινγκ και δεν είναι κάτι το οποίο παρατηρήθηκε μονάχα στη Γερμανία, στη δική μου χώρα. Επομένως πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αποφυγή αυτής της μορφής του ντάμπινγκ Επίσης στο σημείο 32, πέμπτη παρατηρήση λέγεται ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν οδηγήσει σε διάσωση θέσεων εργασίας και υπάρχει μια παραπομπή στις συζητήσεις, ε, θα ήταν να κάνουμε μια παραπομπή στις ε, συζητήσεις των προηγουμένων τριών ημερών, όπου φάνηκε ότι η Κομισιόν θέλει να επιβάλλει εργασία βραχαίως χρόνου στην Γερμανία και επομένως θα πρέπει να υπάρξει κάποια, ε, κάποια αναφορά στο ότι μόνο οι μόνιμες θέσεις εργασίας μπορούν να εξασφαλίσουν την απασχόληση σε συνθήκες κρίσης. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου λοιπόν, εγώ τις έχω διατυπώσει με όσο το δυνατόν πιο επικοδομητικό χαρακτήρα και φυσικά θα τις επαναφέρω και μέσω τροπολογιών. Ευχαριστώ είσαστε πιο συνοπτικοί, σας παρακαλώ, για να δώσω το λόγο ξανά στους προσκεκλημένους μας και έχουμε και άλλο σημείο στη μερίσια διάταξη, ούτως ή άλλως. Κυρία Λίν και μετά κυρία Μάρκη. Ευχαριστώ. Ε, σύντομα σχόλια για τους ομιλητές. Θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Λέτε ότι συχνά ε, κάποιος επιλέγει ελεύθερα την ατυπική μορφή εργασίας. Πόσο συχνά, μπορείτε να μου πείτε. Ε, μιλήσατε για τους φοιτητές, ε, μιλήσατε για διάφορες περιπτώσεις. Επίσης, σε πολλά κράτη-μέλη, πολλές από αυτές τις συμβάσεις ε, σε ορισμένε εργασίε, παραδείγματο χάρη στο consulting κτλ., ε, έχουμε περισσότερες ατυπικές μορφές παρά τυπικέ μορφές εργασία. Επίσης, κάτι άλλο ενδιαφέρον για τη δεδηλωμένη εργασία. Αν ξεφορτωθούμε αυτές τις ατυπικές μορφές εργασίας, ε, θα αυξηθούν οι περιπτώσεις ατυπικής εργασίας ή θα μειωθούν. Κοιτάζω τώρα την έκθεση της κυρίας ε, Γκρινή. Θέλω κάποιες διευκρινήσεις. Στην παράγραφο 4. Μιλάτε για την επέκταση της προστασίας των ε, εργαζομένων που έχουν τέτοιες ατύπικες μορφές εργασίας. Μπορείτε να μου Εξηγήστε τι ακριβώς ε, εννοείτε και τι θέλετε ακριβώς να επιτευχθεί. Στην παράγραφο 7 έχουμε ήδη ε, την ε, νομοθεσία για τα γραφεία βρέσεως εργασίας. πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, σωστά το λέτε. Στην παράγραφο 14, μια διευκρίνηση για τη διατύπωση. Λέτε να εξασφαλιστεί, να εγγυηθεί η ασφάλεια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ε, να εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο εισόδημα. Αυτό εννοείται. Ή, ή ελάχιστο μισθό. Παράγραφος 16. Λέτε ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν εμπιστοσύνη στο εργατικό δυναμικό. Και αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε. Τι ακριβώς εννοείται ότι δεν εμπιστεύονται οι εταιρείε στο εργατικό δυναμικό. Και τελικά στην παράγραφο 18 είναι υπερβολικά έντονη η διατύπωση. Λέτε, καταδικάζει την υπερβολική αντικατάσταση της εργασίας από άτυπες συμβάσεις. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μειώσετε έτσι την, την ένταση αυτής της παραγράφου. Κυρία Μαρκίν, ευχαριστώ. Χάρκιν, συγγνώμη. Ευχαριστώ την εισηγήτρια καταρχήν για την εργασία της και, για τους, και ευχαριστώ και τους ομιλητές. Ένα-δύο σχόλια. Στην παράγραφο 2 μιλάτε για την ανοιχτή μέθοδο ε, συντονισμού που είναι σημαντικό εργαλείο. Ίσως είναι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και ότι δεν ήταν και πολύ αποτελεσματικό αυτό το εργαλείο. μου καταλαβαίνω τι, τι εννοείται. Στην παράγραφο 4 επίσης μιλάτε για διάφορες προτεραιότητες κατά τη μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την υγεία και την ασφάλεια. Ε, γιατί η έκθεση λέει ότι οι εργαζόμενοι με ατυπικές ε, μορφές εργασίας ε, είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους και σε εργατικά ατυχήματα κτλ. Συμφωνώ με αυτό που λέτε στην πράγμα 10 για την έγκαιρη παρέμβαση και μιλάτε για τα δικαιώματα υποστήριξης κατά την περίοδο που χρειάζεται, ούτως ώστε τα άτομα να γίνουν πιο... να έχουν μεγαλύτερη απασχολησιμότητα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η μεταβατική περίοδος γίνεται όλο και μακρύτερη. Έπειτα, συμφωνώ με, την, με τις στρατηγικές διαβίου κατάρτισης, αλλά ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν και στην έκθεση, αν δούμε την έκθεση, είναι ότι οι εργαζόμενοι που έχουν τέτοιε άτυπε μορφέ συμβάσει αποκλείεται ή είναι πιο δύσκολο να εμπλακούν σε τέτοιε προσπάθειε διαβίου κατάρτιση και κατάρτιση. Έπειτα, είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις για αυτά τα θέματα, γιατί αλλάζουν τα πράγματα από κράτο μέλο σε κράτο μέλο και επομένω είναι δύσκολο να έχουμε συνεκτική προσέγγιση. Τώρα, πάλι για αυτέ τι άτυπε μορφέ εργασία. Αυτή η μορφή εργασία δυσκολο να γινουν συγκρίσει για αυτα τα τελευταία χρόνια. Ε, επομένως, δεδομένου αυτού, κάποιες προσαρμογές των δικαιωμάτων των εργαζομένων πρέπει να γίνει για να προσαρμοστούμε σε αυτές τις νέες μορφές. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα συνταξιδοτικά δικαιώματα, με τις εφημερίες, με την αύξηση των μισθών κτλ. Άκουσα αυτά που είπατε για τη Δανία και το ρόλο των συνδικάτων με μεγάλο ενδιαφέρον. Η έκθεση λέει ότι είναι πολύ δύσκολα τα συνδικάτα να δράσουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Ε, επίσης η έκθεση μιλάει για τους εργαζόμενους αυτούς σε άτυπα συμβόλια ε, και λέει ότι συχνά έχουν α, χαμηλό εισόδημα. Ε, μην ξεχνάμε ότι στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020, αν θέλουμε να μειώσουμε το ποσοστό της ανεργίας, που είναι 18%, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με αυτές τις συμβάσεις. Έπειτα, στην έκθεση που λέμε πάλι για αυτούς τους ε, εργαζομένους με ατυπικές μορφές εργασίας, υπερβολικά ατυπικές, λέει ότι τέτοιες καταστάσεις ε, είναι επιζήμιες και για τους εργαζομένους και τους ε, εργοδότες. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον επίσης τα όσα είπαν οι τελευταίοι δύο μιλητές, Business Europe και ο πρόσωπος των κοινωνικών εταίρων και το θέμα της ευέλικης ασφάλειας ε, μας είπαν ότι όταν αυξηθεί η δυνατότητα απασχολησιμότητας, ε, ο κόσμος μπορεί να δράξει τις νέες ευκαιρίες. Αλλά συχνά είναι λίγες αυτές οι ευκαιρίες. Ο εκπροσωπο των κοινωνικών εταίρων είπε ότι Μάλλον υπάρχουν, υπάρχουν κενά μέσα στις δύο περιπτώσεις και η ευελιξία και η ασφάλεια δεν είναι αντιφατικά πράγματα. Το ένα δυναμώνει το άλλο. Μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω ότι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Κλείνω τον κατάλογο των αγοριτών, γιατί έχουμε πέντε ακόμα που θέλουν να λάβουν τον λόγο. Θα ήθελα ο καθένα να μπορέσει να έχει το χρόνο του για να μιλήσει και να κλείσουμε τη συζήτηση. Ε, Κοφερατή και μετά Κορνέλσεν. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. στην πρόταση της ανεφογκρόνης δηλώνει αρχές πολύ σημαντικές που τουλάχιστον στην όλη συζήτησή μας κατά την άποψή μας αποτελούν ένα βήμα σημαντικότατο προς τα εμπρό σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση. Υπάρχουν όμως προβλήματα που δεν οφείλονται σίγουρα στην ε, θέληση της κυρίας Γκρόνιγκ που καθόλου τυχαία τονίστηκαν και θα ήθελα να κάνω μια γενικής φύσεως γρήγορη παρατήρηση, θα δούμε μετά και τις τροπολογίες, αλλά αρκετές φορές άκουσα ότι αυτές οι τυπικές συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές γιατί επιτρέπουν στον κόσμο να διαλέγει. Δεν πιστεύω σε κάτι τέτοιο. Δύο προϋποθέσεις υπάρχουν για μπορεί κανείς να διαλέγει. Πρώτη προϋπόθεση, να γνωρίζει, να διαθέτει γνώση το επίπεδο του μας δείχνουν όμως όλες οι έρευνες ότι η τρομερή πλειοψηφία αυτών των εργασιών δεν έχουν να κάνουν με εξειδικευμένες εργασίες, αλλά λοιπόν ε, όχι κόσμο με σημαντικού υψηλού βαθμού εκπαίδευση, κατάρτιση. Δεύτερη προϋπόθεση που δεν συναντάμε και είναι λεπτότατο στις περιπτώσεις αυτές πρόβλημα. Για να έχει κανείς τα δυνατότητα επιλογής θα πρέπει να έχει προσφορές περισσότερες από, τη ζήτηση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα εργαλεία για όλα αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται με όλα αυτά τώρα εδώ στα πλαίσια της κρίσης. Σημαντικό λοιπόν ένα από τα σημεία που έθεξε η συγγήτρια η κύρωση για όποιον ε, στη θέση της παραδοσικής εργασίας ε, υιοθετεί αυτό το σύστημα ατυπική συμφωνίας όχι για περισσότερη απασχόληση αλλά για μειώσει το κόστος Τη εταιρεία του. Είναι δύο εντελώ διαφορετικά πράγματα, αποκλίνοντα. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε σαν σωστή λογική πράξη και σαν θετική συμπεριφορά. Μάλλον λοιπόν ε, έφτασε η ώρα να επιστρέψουμε σε μία συζήτηση, εδώ θα πω τα πρώτα τη στοιχεία, δεν έχει να κάνει με την έκθεση για την ευελίξη ασφάλεια. Νομίζω ότι ιδιαίτερη σύγχυση δημιουργήθηκε και οι αρχές, εντάξει, τη συμμερίζομαι, Όλες αυτές παραμορφώθηκαν από τη στάση. Εδώ η στάση αυτή είναι αδυναμίας, προβλήματος στην εργασία, όχι ενός λογικού εργαλείου που επιτρέπει να συλλέξει κανείς τα καρπούς, να υποφεληθεί θετικά. Άλλαξε εντελώ ο χαρακτήρας της στάσης. Αυτό από μια μεριά και των αποτελεσμάτων αυτών αποφετέρου. Ορισμένα από αυτά τα θέματα σίγουρα θα πρέπει να τα δούμε και πάλι. Να σας πω ποια είναι. Εντάξει, συμφωνώ, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εμβάθυση. Αλλά εδώ θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα με πρόσβαση και να δούμε ακριβώς και την ε, ε, το ξεκίνημα αυτής της ε, συμφωνίας. Εάν όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με κατάρτιση, όλα αυτά είναι καλή θέληση του εργαζόμενου από τη μεριά ή της επιχείρησης από την άλλη. Δεν ξέρω όμως ε, ιδιαίτερα καλή διάθεση παρόμοιας φύσης. Γιατί αυτή η διαδικασία το να ξεχνωρίζουν αυτά που γνωρίζει ο κόσμος γίνονται από κόσμο που θέλει να χρησιμοποιήσει και στη συνέχεια αυτό τον ε, εργαζόμενο, όχι για κάποιον πρόχειρα έτσι που πάει εκεί εργάζεται και φεύγει, δεν τον προσέχουν ιδιαίτερα. Εδώ λοιπόν ε, δεύτερο θέμα, ο κοινός ενιαίος χαρακτήρας ε, Εάν σε όλες τις χώρες δεν έχουμε αυτό το νέο χαρακτήρα όσον αφορά την αγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ταυτόχρονα αυτό το νέο χαρακτήρα στην κοινωνική του πρόνοια προστασία, αυτές οι ατυπικές συμφωνίες πέρα από τη διάθεση που έχουμε, ίσως ακόμη περισσότερο ξύνουν αυτόν τον χαρακτήρα, ένα μέσο περιορισμένο και να χρησιμοποιηθεί κυρίως αν ε, δεν υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα για όποιον ε, δέχεται ένα παρόμοιο ε, συμβόλαιο ή όπως τον άλλον. Αυτό σημαίνει μια μείωση του κόστους, γιατί και τα δικαιώματα σημαίνουν ένα κόστος. Σημαίνει ότι η επιχείρηση θα στραφεί προς τα εκεί για την ίδια διάρκεια εργασίας να δώσει σε πολλούς συμβόλαια παρόμοια τυπικά. Το ίδιο και για την κοινωνική προστασία και εδώ για τους πιο νέους. Αυτή η επανοβανόμενη και διαδεμένη χρήση ...παρομοίων συμβολέων σε αυτές τις συμφωνίες, στην νομοθεσία πολλών χωρών, τι σημαίνουν. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για όταν προχωρήσει ηλικία και τι θα γίνει όταν ε, ε, πάει, βγει από την αγορά εργασίας. Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την κοινωνική προστασία και θα έχουμε κόσμο που θα έχει ε, τη διάρκεια συμβόλαιο και εντάξει μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση και από την άλλη μεριά κόσμο που για τα ίδια, την ίδια διάρκεια θα εργάζονται, αλλά επειδή συνεχώς θα ανατεώνουν αυτά τις ατομικέ συμβάσεις, η προστασία τους θα είναι περιορισμένη. Τώρα να σας πω ότι σημερινά οι νέοι, όταν κατανοήσουν αυτή τη διαφορά, ίσως θα είχαν και μια στάση διαφορετική που να μην ε, προχωρούν προς μια κοινωνική συνοχή. Και ακόμα ένας τίτλος, ο κοινωνικός διάλογος. Να σας πω ότι με την ίδια είμαι απόλυτα σύμφωνο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εκπροσώπηση που έχει να κάνει με τις δικαλικέ οργανώσει, αλλά και με τις ε, ενό εργοδοτών. Είναι εκπρόσωπο έτσι αυτής της ε, και με την άλλη εργασία την ε, διαδομένη που είναι ορατή για να ισχυθεί αυτό ο κοινωνικό διάλογο θα πρέπει να υπάρχουν και εργαλεία που να βοηθήσουν την όλη οργάνωση την καλή. Κορνέλσεν και Φιγκερέντο, σας παρακαλώ τώρα να είσαστε όσο το δυνατόν σύντομότερες. Κορνέλσεν. Ευχαριστώ. Οι ατυπικές σχέσεις εργασίας σημαίνουν ότι πρέπει να υπάρχουν και τυπικές σχέσεις εργασίας. Να υπάρξει λοιπόν μια πραγματική στην περίπτωση των γυναικών μια πραγματική κατανομή μεταξύ των ε, ευθυνών στον οικοκυριό και ευθυνών στο χώρο εργασίας. Επομένως, η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα είναι να υπάρξει συμφιλίωση του χώρου εργασίας και του οικιακού χώρου. Όλοι οι άντρες και οι γυναίκες οι οποίοι θα μπορούν να εργάζονται, θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται, αλλά σημαίνει αυτό ότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία θα πρέπει να τα φροντίσουμε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν με μερική απασχόληση ή με ευελίκτες ώρες, αυτό μπορεί να ευνοήσει μια καλύτερη κατανομή του βάρους αυτού. Αν υπάρχουν δύο σύντροφοι οι οποίοι δουλεύουν τρεις μέρες τη βδομάδα ο καθένας, αυτό είναι μια μέρα παραπάνω από ένα άτομο που δουλεύει πέντε μέρε τη βδομάδα και αυτό δίνει περισσότερο χρόνο για να φροντίζουν τα παιδιά και οι ηλικιωμένου γονεί. Για μένα λοιπόν οι δυνατότητε αυτέ για του εργαζομένου, όσο πιο πολλέ είναι οι εύκαμπτε μορφέ εργασία, τόσο το καλύτερο. Βέβαια, πολλέ φορέ η ευελιξία χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα εκμετάλλευση των εργαζομένων. Επομένω, εμεί ω πολιτικοί έχουμε το καθήκον να προστατεύσουμε του εργαζομένου όσο μπορούμε περισσότερο, ενώ συγχρόνω του δίνουμε το ευρύτερο δυνατό φάσμα ευελιξία. Όπως και η κυρία Λίν, εγώ θα ήθελα να ακούσω τις προτάσεις των ομιλητών για την παροχή αυτής της προστασίας που ανέφερα. κυρία Φιγκερέντο και ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φιγκερέντο. Ξέρω ότι αυτά τα ερωτήματα για τις ατυπικές σχέσεις εργασίας, για την ασφάλεια, την ευελιξία, όλα αυτά, δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω όμως ότι για τη χώρα που ξέρω καλύτερα, τη δική μου χώρα, την Πορτογαλία, ο πολλαπλασιασμός των θέσεων ατυπικής εργασίας, των μη συμβατικών μορφών εργασιακής σχέσης, συνδέεται ιδιαίτερα με την ευελιξία της εργασίας, την αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, ιδίως στον τομέα των κατασκευαστικό, και μια υποβάθμιση της αξίας εργασίας, ιδίως της εργασίας των νέων και των γυναικών, που τώρα πια πολύ σπάνια μπορούν να πετύχουν μια πραγματική θέση εργασίας. Το λέμε αυτό ευέλεξε ασφάλεια. Ωραία. Στη χώρα μου οι περισσότεροι ε, εργαζόμενοι λένε δεν τη θέλουμε χάρισμά σα η ευέλικτη ασφάλεια. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι εργασία με δικαιώματα. Θέλουμε εργασία η οποία να αναγνωρίζεται, η οποία να αναγνωρίζει την προσπάθειά μας και τον κόπο μας και να μας δίνει αποδοχές αξιοπρεπής, όχι αποδοχές αθλειότητας και ένδυας. Αποδοχές μας δίνουν τη δυνατότητα να ζήσουμε με μια αλλάξη αξιοπρέπεια που σέβεται την εργασία των γυναικών και των ανδρών. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο συμβαίνει έχει αυξηθεί με εκθετικό τρόπο η μορφή αυτή εργασίας, οι μη συμβατικέ μορφές εργασίας, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία της ευέλικης ασφάλειας. Με εκθετικό τρόπο έχει αυξηθεί η ατυπική εργασία, η μη συμβατική εργασία. Και αυτό οδήγησε σε μία επιδίνωση των συνδικών εργασίας και σε μία υποβάθμιση της αξίας της εργασίας. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς θα απαντηθούν αυτά τα θέματα. Και φυσικά υπήρξε και αύξηση της ανεργίας. Γιατί υπάρχει και μια άλλη κατάσταση, την οποία με σοκάρει εμένα, ιδιαίτερα στο σημείο 10 λέει η συγγήτρια, ότι το πιο σημαντικό για την ε, απασχόληση είναι να υπάρχει μια θέση εργασία. Α υπάρχουν θέσει εργασία ακόμα και αν επισφαλεί. Όχι, για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορώ να δεχτώ μια τέτοια αντιμετώπιση ότι χρησιμοποιείται η αύξηση της ανεργίας ώστε να είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι να δεχτούν ό,τι να είναι σε επίπεδο εργασίας, ακόμα και ανεπισφαλής. Ευχαριστώ. Το Μασμά, Ελιζαμπέτ Μωρά, μετά εγώ. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε και τον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι έχουν ε, σημειώσει ότι είναι θαυμάσια η έκθεση της κυρίας Γκρίνη, η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εμείς φυσικά θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε με τις τροπολογίες μας και με τις προτάσεις μας. Ο κύριος ε, Χέντελ έφυγε, αλλά είπε ότι θα ξαναέρθει. Στο σημείο 4 αναφέρεται ότι πρέπει να μπορούμε να φτάσουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ευελιξίας. Στην έκθεση Κίσεν επίσης αναφέρεται ότι θα μπορέσει να υπάρξει και συμβιβασμό τη εργασίας με τον οικογενειακό χώρο. Λοιπόν, πιστεύω ότι όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας. Αγαπητέ κύριε Χέντελ, είπατε ότι δεν συμφωνείτε με το σημείο 29 να ζητηθούν οι... να ζητηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν αυτοί όλο το βάρος. Εγώ νομίζω ότι στη Γερμανία έχουμε αυτή την παράδοση το να εξασφαλίζουμε το ότι όταν υπάρχουν ατυπικέ θέσει εργασία υπάρχουν και οι απαραίτητε διασφαλίσει. Προ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι πολλέ φορέ οι ατυπικέ σχέσει εργασία έχουν μεταμορφωθεί σε τυπικέ σχέσει εργασία. Και για την Πασκάλ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο σημείο 19 επίση είναι σαφέ ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό με κοινό τρόπο, να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει. Έχουν διαφορετικό κέντρο βάρου οι εθνικέ πολιτικέ. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια κοινή ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία να υποστηρίζει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Για μένα αυτό είναι απόλυτα ορθό. Στο σημείο 29 και πάλι σα λέω ότι θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρξουν έγκαιρε επενδύσει, Γιατί πάντα δράμε πυροσβεστικά, παραδείγματο χάρη με το Ευρωπαϊκό Ταμείο παγκοσμιοποίηση, Αλλά αυτό μπορεί να είναι μονάχα ένα κομμάτι τη όλη εργασία μα ή το θέμα των μικροποστώσεων. Πολλές φορές δεν είναι τα μέτρα τα οποία εμείς διαλέγουμε, αυτά τα οποία θα μπορούν να παίξουν ένα προληπτικό χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο και να ξεδιπλώσουμε την φαντασία μας, ώστε να μπορούμε να έχουμε μέτρα τα οποία θα δρουν έγκαιρα και προληπτικά. Και πιστεύω ότι δεν ξέρω αν έχω αντιμετωπίσει όλα τα σημεία κριτική που ήταν πολλέ φορέ οξύ, αλλά νομίζω και η Πασκάλ Γκρινή θα μπορέσει να απαντήσει από τη δική τη πλευρά. Κυρία Μωρά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Την Γκρίνιγκ θα ήθελα να την ευχαριστήσω γιατί συνέταξε μια παρόμοια έκθεση δύσκολη με πολλά στοιχεία έχει να κάνει και με ευαίσθητο θέμα, κάτι που εξελίσσεται συνεχώς και ταυτόχρονα ταυτόχρονα στα πλαίσια μέσα στο κέντρο του κυκλώνα αυτή τη κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Να επιμείνω σε τρία σημεία πάνω. Το πρώτο παλό έχει να κάνει με τις άτυπε άτυπες συμβάσεις. Ε, επειδή ακούσαμε πολλά και διάφορα στην έκθεση αυτή. Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε ορισμένες περιπτώσεις ε, που έχουν να κάνουν με νέα μορφή οργάνωση εργασίας που είναι σύνολα εργοδοτών ε, που δεν εμφανίζονται εδώ, αλλά είναι κάτι το θετικό που θα μπορούσε να γίνει. Είναι μια νέα μορφή άτυπη σύμβασης και εδώ στην παράγραφο 5 και 17 διάφορες προσθήκες που θα μπορούσαμε να έχουμε για αυτά τα σύνολα εργοδοτών, ομάδες εργοδοτών και διευκρινήσεις για την ε, εργασία που δεν είναι κανείς φυσικά, δεν παρίσταται φυσικά και έχουν να κάνουμε όλα αυτά και με την υγεία στο δικαίωμα συνεχού κατάρτιση πολλά και διάφορα για αυτά τα δύο στοιχεία, τα δύο θέματα που είναι καινούργια στην όλη οργάνωση εργασίας, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένε συντηρηματικέ διευκρινήσει. Δεύτερο σημείο για την ευελίξη ασφάλεια και για την σίγουρη επαγγελματική πόρια θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα. Όπως η κυρία Ακίν το είπε πριν από λίγο. Να πούμε ότι χρειάζεται να επιβραβεύεται η πρώτερη με μια πανακατάρτιση αν γίνεται και με μια απασχόληση ε, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής ακριβώς ε, αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζει αυτές τις συμβάσεις. Ε, όχι τη στιγμή που αντιμετωπίζει κολλίες με απολύσεις, όχι τότε να λέει να επικυρώνει αυτό το μπλούτο προϊόντων και να προσπαθεί να επανακαταρτήσει καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της ζωής τους. Όλα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται, θα πρέπει να αναπτύσσονται, τα προσόντα αυτά δηλαδή μέσω της κατάρτισης αυτής. Για το πρόβλημα αυτό της ευελίξης ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτά θα ήθελα να είμαστε περισσότερο συγκεκριμένοι για τις συμφωνίες που χωρίς ε, εξειδίκευση προέρχονται από μια κατάρτιση. Είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη ομάδα να αντιμετωπιστεί αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα πούμε έτσι με μια φρασούλα σε αυτά τα πλαίσια. Χρειάζεται όμως ειδική στρατηγική. Για να τελειώνω κύριε Πρόεδρε, για τις νέες μοσφές ε, κοινωνικού διαλόγου είδαμε πολλά να γράφονται αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται μια, ένας επαναπροσδιορισμός πραγμάτων σχετικά με το διαφορετικό αυτό χαρακτήρα στις επιχειρήσεις κοινωνικού διαλόγου. Τι βλέπουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο κοινωνικός διάλογος δεν έχει την ίδια μορφή όπως τις μεγάλες εταιρείε. Δεν προστατεύεται, δεν υπάρχει η ίδια παρότρινση με τον ίδιο τρόπο δηλαδή. Χρειάζεται αυτό να το δούμε διεξοδικότερα, να δούμε τη διαφοροποίηση αυτού του κοινωνικού διαλόγου ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Επίσης κάτι να προσθέσω, ότι στα πλαίσια αυτών των ε, διαφορετικών συμβάσεων ε, θα πρέπει να δούμε τη διαφοροποίηση και την όλη οργάνωση σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή αυτών των επιχειρήσεων. Και γνωρίζετε κάτι ειδικά ότι υπάρχει εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας ανάμεσα στην, ε, σε γεωργικό χώρο και σε αστικό χώρο. Υπάρχουν ε, στην Ήπεθρο εταιρείε επιχειρήσεις. Το πρόβλημα δεν ε, τίθεται εκεί με τον ίδιο τρόπο, αλλά μερικές φορές ακόμα δυσκολότερο είναι εκεί να λυθούν τα προβλήματα. Για να τα δούμε λοιπόν αυτά, να τα εξετάσουμε επίσης, αυτόν τον, εξετάσουμε αυτόν τον διαφορετικό χαρακτήρα. Και σας ευχαριστώ που με αφήσατε να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιε ερωτήσει προ την εισηγήτρια και του ομιλητέ μα, κυρίω τον κύριο Ντεκαγιό, για το θέμα τη εξασφάλιση τη επαγγελματική πορεία. Γιατί ένα από του λόγου που υπάρχει αυτή η έκθεση είναι να αναπτύξουμε αυτή την ιδέα. Αλλά δεν υπάρχει τελικά τίποτα για αυτό, για αυτή την ιδέα. Τίποτα, τίποτα πραγματικά. Η ιδέα ευέλικτη ασφάλεια και ασφάλεια τη επαγγελματική πορεία ε, τελικά ταυτίζονται. Δηλαδή το δεύτερο αφορά το πρώτο. Αυτέ όμω οι δύο έννοιε είναι τελείω διαφορετικέ. Πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ευελιξασφάλεια και εξασφάλιση τη κοινωνικής, της επαγγελματικής συγγνώμη, πορεία. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε για τι νέε μορφέ εργασία, για τι άτυπε μορφέ εργασία, μόνο, θα, μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν εξασφαλίσουμε την επαγγελματική πορεία των εργαζομένων. Και ελπίζω στη συνέχεια αυτή τη συζήτηση μέσω των τροπολογιών κυρίω να δώσουμε απαντήσεις και σε αυτό το τομέα. Ζητώ συγγνώμη που θα είμαι τόσο αυστηρή με το χρόνο που θα δώσω στο, στον καθένα από εσά, που θα είναι μόνο δύο λεπτά. Δεν έχω παραπάνω. Ελπίζω να έχουμε το χρόνο αργότερα στα πλαίσια της εκπόνησης αυτής της έκθεσης να τα ξαναπούμε με μεγαλύτερη ησυχία. Αλλά θέλω να δώσω και σε εσά το λόγο και στην εισηγήτρια και έχουμε ακόμα ένα σημείο στη μερίσια διάταξη. Λοιπόν, θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπιλέτα ε, και θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι ομιλητέ με την σειρά που μίλησαν ε, προηγουμένω. Κυρία Μπιλέτα, να απαντήσω σε μία ερώτηση για το πόσο υψηλά πρικισμένοι εργαζόμενοι έχουν τέτοιες άτυπες μορφές εργασίας. Σε μία από τις μελέτες μας λέμε ότι το 8% ε, των ανθρώπων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τέτοιες πολύ ατυπικές μορφές εργασίας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι πόσο καιρό μένει κανείς σε τέτοιου είδους υπερβολικά ατυπικές μορφές ε, και πόσο πολύ μπορεί να κινηθεί από τις υπερβολικά ατυπικές μορφές σε άλλες μορφές, που δεν είναι ίσως εντελώς μόνιμες, αλλά που είναι κάποιες μορφές που σου δίνουν περισσότερα δικαιώματα, κυρίως συνταξιδοτικά δικαιώματα, σε περισσότερα δικαιώματα σε επίπεδο υγειονομικής κάλυψης κτλ. Αυτό νομίζω είναι το βασικό πρόβλημα. Η μετάβαση από την υπερβολικά άτυπη μορφή εργασίας Προ μια άλλη μορφή εργασία είναι πολύ πιο γρήγορη για αυτού που έχουν πολλά προσόντα και πολύ αργότερη για αυτού που έχουν λιγότερα. Μία άλλη ερώτηση αφορούσε τι γυναίκε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε ε, για τη διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλλα που υπάρχει. Έχουμε πολύ λίγα δεδομένα ποσοτικά για αυτή τη διάκριση. Παραδείγματο χάρη έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι στο Λουξεμβούργο το 99% των εργαζομένων που δουλεύουν λιγότερο από 10 ώρες, το 99% είναι γυναίκες. Είναι ένα παράδειγμα, έτσι. Είναι ένα στοιχείο όμως. Αλλά υπάρχουν υπερβολικά πολλές γυναίκες σε αυτές τις πολύ άτυπες μορφές εργασίας. Και φυσικά αυτό έχει επίπτωση στην ασφάλεια την επαγγελματική τους στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να τονίσω τρία ή και τέσσερα σημεία. Πρώτα απ' όλα, από Αντώνα στην Τεκαγιό, είναι πολύ θετικό αυτό που θέσατε σαν ερώτημα, τι ακριβώς κάνουμε στον τομέα αυτό και αναφερθήκατε στην έρευνα της αγοράς. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε εκπονήσει είναι ένα πολύ καλό, καλή βάση για την υπεραιτέρω ανάπτυξη των δράσεων μας σε εθνικό επίπεδο και θέλω να καλωσορίσω αυτή τη μνήμα που κάνατε πώς θα δημιουργήσουμε την έννοια της προστασίας για τους εργαζομένους ή πώς θα γίνει αυτό. Το έθεσε το ερώτημα κυρία Κονέλσεν, αν δεν απατώμε. Θέλω να τονίσω ότι η ευελιξή ασφάλεια αφορά και την ασφάλεια και την ευελιξία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό. Δεύτερον, <clears throat> εμείς ως κοινωνική εταίρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε συμφωνήσει πολλές φορές το 1997-1999 σε μια σειρά συμφωνίες που έγιναν μετά οδηγίες για εργασία συγκεκριμένου χρόνου και εργασία ε, μερικού, μερικής απασχόλησης και αναφέρθηκε και το θέμα της τηλεεργασίας σχετικά που ανέφεραν πολλοί ομιλητέ. Ο στόχος αυτών των συμφωνιών ήταν να τεθεί σε εφαρμογή η αρχή της μη διάκρισης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ήδη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά και επομένως η δράση τώρα θα πρέπει να αναλυφθεί σε εθνικό επίπεδο. Μια τελευταία παρατήρηση για το θέμα της γκρίζα ή μαύρης οικονομίας. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτός είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες και εμείς χαιρετίζουμε αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσης για την πλευρά αυτής της οικονομίας γιατί αυτοί που είναι στην ε, παραοικονομία είναι οι πραγματικά απόκληροι της αγοράς εργασίας και δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία σύγχυση με μορφές εργασίας οι οποίες είναι νόμιμες και όταν μιλάμε για εφαρμογή του νόμου σας λέω ότι η ευέλικτη εργασία είναι νόμιμη και παγιωμένη. Σας ευχαριστώ. Ναι, αλλά είναι και μερικές φορές επισφαλής. Δεκαγιών δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Εντάξει, επιβεβαιώνω. Έχουμε τι 45 σελίδες στα αγγλικά αυτή την ανάλυση για να δούμε αυτό το περίπλοκο χαρακτήρα του προβλήματος. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε σαν την γκρέμα, σαν τη γη στο παγωτό απάνω σε όλα τα θέματα, αλλά είναι η μορφή αυτή ιδιαίτερα περίπλοκη. Αν θέλουμε μια σοβαρή συζήτηση στην Ευρώπη και επικοδομητική, θα πρέπει να δεχτούμε αυτόν τον περίπλοκο χαρακτήρα του ε, αυτού του ευελίξη ασφάλεια και να αποφεληθούμε από όλα και όχι να το βάζουμε παντού σαν σάλθα, σαν μαϊντανό που πάει παντού. Εδώ λοιπόν ε, δεύτερο στοιχείο, δύο ακόμα εκθέσει. Ε, το είπε ο συνάδελφο εδώ, Παρακαλώ για το εργαλείο αυτό το 29 σημείο εμείς ευρωπαϊκό επίπεδο σαν κοινωνική εταίρη, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ε, και θα πρέπει να δούμε άλλη μια συμφωνία. Είχαμε τρεις συμφωνίες έτσι για να πω καταλέξω ότι γίνεται στα πλαίσια τα ευρωπαϊκά ένα πρόγραμμα δράσης για ατυπά ε, τυπικά προσόντα. Υπάρχουν λοιπόν εδώ με του κοινωνικούς εταίρους τι σημαίνει αυτή η επικύρωση εισαγωγικά είναι κάτι πολύ σημαντικό σε εκείνου που αντιμετωπίζουν αυτήν την επισφαλή εργασία σε άτυπε συμβάσει. Ή έστω και χωρί αυτέ. Τι κάνω όλοι αυτοί, είναι ή έστω και χωρι αυτε Τι κάνουν όλοι αυτοί. Είναι ισχνη κατάρτισης και να Σω αυτού που έχουν διαλέξει άλλη μόρφη, το λέει και η παροιμία, υπάρχουν ε, και ψάρια που πετάνε, αλλά δεν είναι ο κανόνα αυτό. Εδώ τα περισσότερα είναι χωρί ιδιαίτερη κατάρτιση αυτέ οι άτυπε συμβάσει. Ε, έχουν κατάρτιση, δεν έχουν αναγνώριση των προσόντων του. έστω και αυτά που έχουν αποκτήσει με αυτές μη κατάλληλε κατάρτιση. Ε, αν δούμε όμω, υπάρχει και αναγνώριση κοινωνική το θέμα αυτό. Τρομερή προσπάθεια πρέπει να γίνει σε αυτή την κατάρτισή του και αναγνώριση αυτών των προσόντων Τώρα, θέλουμε να εργαστούμε λοιπόν ε, για αυτή τις άτυπες συμβάσει και επανενταχθούν ακριβώς ε, σε αυτή τη μορφή εργασίες ε, αόριστης διάρκειας, εδώ θα πρέπει να δούμε ότι αυτοί που φαλάζουν είναι λιγότερο εκπαιδευμένοι και με περισσότερη επισφαλή θέση. Και έχουμε και πάνω από τους 50 ετών. Όταν βλέπουμε αυτό το θέμα, το θέμα γενικά είναι τρομερή αντίφαση εκεί και όλοι συμφωνούμε για αυτή την κατάρτιση, αλλά τα πρώτα χρήματα που θυσιάζονται είναι η επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Δεν φτάνει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχουν τα πράγματα, αλλά μετά τη γίνεται εφαρμογή του που είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Ευχαριστώ. Μιλήσαμε για την εξασφάλιση της επαγγελματικής καριέρας, ίσως θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Κάποτε θα πρέπει να μπούμε και σε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Κρίνου, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο διαμακρόν σήμερα, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και την έκθεση ΣΕΡΚΑ στη συνέχεια. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Έχετε το λόγο με μεγάλη συντομία. Για τους συναδέλφους πάντα θα υπάρχει η ευκαιρία να καταθέσουν τροπολογίες μέχρι το τέλος Μαρτίου. Αυτό το οποίο εγώ ήθελα να πω είναι να αναφερθώ σε δύο ερωτήματα τα οποία κατατάθηκαν. Για μένα η θέση, η σύμβαση αορίστου χρόνου με σταθερή θέση εργασίας είναι ο κανόνας, ενώ οι ατυπικές συμβάσεις είναι κάτι το περιθωριακό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι υπάρχουν γυναίκε οι οποίε προτιμούν να μην εργάζονται με πλήρη απασχόληση γιατί θέλουν να συμβιβάσουν την οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ζωή. Αυτό όμω δεν είναι κανόνα. Αυτό είναι μια εξαίρεση που αφορά μονάχα ορισμένα άτομα. Δυστυχώ οι ατυπικέ σχέσει εργασία δεν είναι αντικείμενο επιλογή αλλά επιβολή τι περισσότερε φορέ. Επίση για τα διάφορα ερωτήματα εγώ κατέγραψα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, την κατάρτισή τους και όλα αυτά. Για μένα όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν αντικείμενο, αποτελούν μάλλον κομμάτι των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τη μορφή σύμβασης που έχουν. Και πιστεύω ότι με την έργαση αυτή πρέπει να έχουμε μια τέτοια οπτική γωνία και να ζητήσουμε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν ακριβώς να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων ανεξάρτητα από τη μορφή εργασία. Στην παράγραφο 10 η κυρία Φιγκερέντο αναφέρθηκε και εκεί δεν είπα ότι θα πρέπει να είναι η ατυπική εργασία η απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά κάνω την διαπίστωση ότι τα άτομα τα οποία μένουν άνεργα για πολύ καιρό έχουν μετά τεράστιες δυσκολίες για να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Επομένως, αν μπορούν να έχουν πολύ γρήγορα μια θέση εργασίας, ίσως περιορισμένη στο χρόνο ή με μερική απασχόληση, τουλάχιστον κρατάνε ένα πόδι στον χώρο της εργασίας και αυτό τους διευκολύνει στη συνέχεια να βρουν μια κανονική θέση εργασίας. Αυτό ήθελα να πω εδώ, στο σημείο 10. Επίσης, κυρία Λίν, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην αγορά εργασίας, αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν κάποια μεγάλη ορατότητα σε σχέση με το τι θα γίνει στο μέλλον. Θα πρέπει εκεί πέρα να προσαρμόσουν τις ανάγκες τους στις ε, μορφές θέσεων εργασίας. Και εδώ για αυτό το λόγο εγώ ανέφερα ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια κύρωση αν μεταμορφώνονται οι κανονικές θέσεις εργασίας σε ατυπικές θέσεις εργασίας. Πρέπει να είμαστε αυστηροί στο θέμα αυτό η εξασφάλιση της επαγγελματικής καριέρας, εγώ το έχω αναφέρει, δεν υπάρχει μια ειδική παράγραφο στην έκθεση, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια, αλλά δεν είμαι καθόλου κλειστή για μια τέτοια μνήμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει σε όλο το μήκος της έκθεσης. Ο στόχος μου είναι πραγματικά να υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός εργαζομένων σε φυσιολογικές τυπικές σχέσεις εργασίες. Λυπάμαι δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους, αλλά προσπάθω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Δεκή Πρόεδρος. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε έτσι μία πρώτη εξέταση αυτή της έκθεσης. Και Έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες, έτσι σφιχτή, 29 Μαρτίου μέχρι το μεσημέρι. Και μετά, στις 27 Απριλίου θα τις α, συζητήσουμε και η υιοθέτηση 2 Ιουνίου. Πάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Αλεχάνδρου Σέρκας. Είναι μια έκθεση που αφορά την ενιαία διαδικασία αίτησης για διαμονή και εργασίας. Είναι παλιό θέμα και η καθήλια αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή ε, Δημοσίων Ελευθεριών. Ο εισηγητής θα μας εξηγήσει το θέμα αυτό και πού φτάσαμε με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν σταματήσει και ξανάρχισαν. Merci. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως πράγματι είπατε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει κάποιο ιστορικό ήδη και πρέπει να γράψουμε κάτι σε ένα φύλλο χαρτί και να μην το αφήσουμε κενό, αλλά μόνο σε μία σελίδα. Ξεκινήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση το 2008 με μία έκθεση της Επιτροπής μας που πήγε στην ε, Ολομέλεια στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή είμαστε μονάχα, τότε είμαστε μονάχα σε φάση διαβούλευση, αλλά με βάση της νέας διαδικασίας έχουμε πλήρη συναπόφαση. Είναι μακρά η ιστορία της προσπάθειας ρύθμισης των συνδικών εργασίας των ε, υπηκών τρίτων χωρών που βρίσκονται με νόμιμο τρόπο στην Ευρώπη. Μιλάμε για την νόμιμη μετανάστευση. Υπήρξε ένα μακρό ιστορικό στο Κοινοβούλιο, στη Κομισιόν, αλλά και στο Συμβούλιο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι αυτή είναι μια υπόθεση στην οποία είμαστε συναρμόδια με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Δεν είμαστε απόλυτα αρμόδιοι παρά μόνο για ορισμένα από τα άρθρα του σχεδίου οδηγίας, όχι για το σύνολο της οδηγίας. Γι' αυτό η έκθεσή μου περιορίζεται σε αυτά τα άρθρα και στις αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις. Η ιστορία αυτού του θέματος είναι αρκετά γνωστή. Η μετανάστευση τώρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα υπήρξε ένα θέμα που ενδιαφέρει μάλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση και απλώς για να σας υπενθυμίσω ορισμένα από τα βασικά κεφάλαια αυτού του θέματος, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μετά από την έγκριση συνθήκης Λισαβόνας υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις κομισιών σε σχέση με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την νόμιμη μεν και την παράνομη δε μετανάστευση το Σύμβουλο πάντα είπε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί με την παράνομη μετανάστευση, αλλά για όλους αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη για να έχουν μια καλύτερη ζωή για την, ε, τον εαυτό τους και της οικογένειάς τους, αλλά για να βοηθήσουν και την Ευρώπη στην οικονομική ανάπτυξή της και τη διατήρηση του κοινωνικού μοντέλου τους, οι εργαζόμενοι αυτοί που είναι νομίμως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς έχουμε δεσμευτεί σταδιακά να άρουμε όλους τους φραγμούς που εμποδίσουν την επίτευξη της αξιοπρέπειάς τους ως ατόμων και την δυνατότητά τους να απολαμβάνουν πλήρως του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν της απόλυτης ισότητος μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων στα από τα κράτη-μέλη μας και των μεταναστών νομίμων εργαζομένων. Θέλω να σας πω ότι αυτή η οδηγία όπως και όλες οι, όλα τα στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας σέβονται την αρχή της επικουρικότητας. Δεν μιλάμε για τα δικαιώματα στην εργασία ή και τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά είναι θέματα τα οποία ρυθμίζονται από κάθε κράτος βάσει του δικού του θετικού δικαίου. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ είναι το να μπορεί ο μετανάστης εργαζόμενος στο οποιοδήποτε κράτος μέλος να απολαμβάνει ίσων δικαιωμάτων με τον ε, εθνικό εργαζόμενο παρά το γεγονός ότι δεν έχει το ίδιο νομικό καθεστώς, την ίδια νομική ιδιότητα. Μιλάμε λοιπόν για την ισότητα και όχι για το συγκεκριμένο περιεχόμενο με το οποίο θα επενδύσει το κράτος μέλος αυτά τα δικαιώματα. Αυτά λοιπόν αναφερόντουσαν σε μία οδηγία του, σε μια ανακοίνωση του 2005 μετά την έγκριση συνθήκης Λισαβόνας. Ο στόχος ήταν να γίνει πιο ελκυστική η εργασία στην Ευρώπη για τους νόμιμους εργαζόμενους. Μετά από την οδηγία αυτή του 2000, την ανακοίνωση του 2005 υπήρξαν και άλλες ανακοινώσεις που ανέφεραν ότι συνδέεται το θέμα τη νομή μετανάστευση με την κοινωνική ενσωμάτωση των εργαζομένων και δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ενσωμάτωση χωρί ισότητα στον εργασιακό τομέα. Και σήμερα έχουμε τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που αναφέρεται έστω και συνοπτικά στο άρθρο 12 που λέει ότι για όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη και ακόμα για τους πολίτες τρίτων χωρών υπάρχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, υπάρχει το δικαίωμα της παιδείας, το δικαίωμα της ισότητας σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και στο άρθρο 21 αναφέρεται η μη διάκριση, το δικαίωμα των υπηρεσιών ε, που έχουν να κάνουν με την εγκατάστασή τους τι δίκαιε συνδίκε εργασία επίση, στο σημείο 34 αναφέρεται η κοινωνική ασφάλεια, στο άρθρο 35 είναι η προστασία τη Υγεία των εργαζομένων. Πρέπει εμεί λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να δώσουμε το ερώτημα. Αυτά τα δικαιώματα που έχουν οι ηθαγενεί ενό κράτου μέλου. Είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε σε όλου αυτού οι οποίοι είναι νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το πράξουμε αυτό χωρί κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση θα πρέπει να απαντηθεί από την ε, Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Θα πρέπει να αποφασίσει αν πρέπει να δοθεί αυτή η ισότητα σε όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσει για αυτούς οι οποίοι είναι εποχιακά εργαζόμενοι, για αυτούς για τους οποίους ε, εκκρεμεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε ποιε είναι οι εξαιρέσει στο δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημοσίου Ελευθεριών. Αυτοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν λοιπόν την ισορροπία σε σχέση με το ποιε θα είναι ομάδες των μεταναστών που θα πρέπει να προστατευτούν από αυτήν την ισότητα. Εμείς όμως θα πρέπει να σταθούμε σαν Επιτροπή Απασχόλησης στο άρθρο 12. Δηλαδή όλα αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να ισχύουν για τους μεταναστές εργαζομένους ή θα εξαιρέσουμε ορισμένα και θα επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να αφαιρέσουν ορισμένα δικαιώματα τα οποία ισχύουν για τους ηθαγενείς τους και επομένως θα τα αρνηθούμε αυτά τα δικαιώματα στους εργαζόμενους τρίτων χωρών που έχουν το δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τροπολογίες που έλαβα αγαπητοί συνάδελφοι νομίζω ότι έχουν σε στόχο να βελτιώσουν το κείμενο της Κομισιόν γιατί το κείμενο της Κομισιόν που είναι ένα θετικό κείμενο που σίγουρα βελτιώνει την τωρινή κατάσταση περιλαμβάνει και ορισμένες ασυνέχειες και ασυνέπειες οι οποίες δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν και που θα τεθούν εν αμφιβόλο αυτές οι απόψεις από την κοινωνία των πολιτών, από τα συνδικάτα κτλ. Θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα δώσουμε απάντηση σε αυτά τα ερώτηματα. Τέσσερις τροπολογίες που είναι πιο σημαντικές είναι αυτές τις οποίες θα αναφερθώ. Γιατί κατά την άποψή μου φύγουν ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα και θα πρέπει να είναι και αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο για να επιληθούν τα θέματα αυτά. Οι τροπολογίες αυτές είναι... Αρχίζω από τα πιο σημαντικά η 13 καταρχήν. Στο άρθρο 12 της πρώτας οδηγίας η Κομισιόν δίνει την έγκριση στα κράτη-μέλη να αφαιρέσουν το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλειας με την εξαίρεση του επιδόματος ανεργίας από τους μετανάστες εργαζόμενους. Δηλαδή μπορεί ένα κράτος μέλος να πει ότι δεν μπορεί να έχει υγειονομική προστασία ή στεγαστικά στεγαστική υποστήριξη, υποστασία της οικογένειας ένας μετανάστης εργαζόμενος. Αυτό νομίζω ότι ανατρέπει όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, ισότητα δικαιωμάτων για ένα θέμα το οποίο είναι κεντρικό για την ευρωπαϊκή ε, κοινωνία. Ρώτησα λοιπόν την Κομισιόν και το Συμβούλιο γιατί να χάνει αυτά τα δικαιώματα για την υγειονομική περίθαλψη ένα μετανάστη. Ποια είναι η επιχειρηματολογία πάνω στην οποία εδράζεται κάτι τέτοιο, μια τέτοια εξαίρεση. Εφόσον πρόκειται για άτομα τα οποία νομίμως βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμένα μου φαίνεται λοιπόν ότι αυτό δεν ε, θα ήταν ορθό. Η τροπολογία 12 αφορά και πάλι τον εργαζόμενο ο οποίος χάνει τη θέση εργασίας του. Και θα πρέπει εδώ να υπάρχει η προστασία από την πλευρά της ε, Κομισιόν να αποδεχτεί το γεγονός ότι κάποιος ο οποίος χάνει τη θέση εργασίας του δεν πρέπει να χάσει το δικαίωμα να συνεχίσει να είναι μέλος μιας εργατικής ένωσης ή κάποιας ένωσης μεταναστών. Αυτό είναι μια αβάσιμη και αστήριχτη εξαίρεση την οποία δεν πρέπει να δεχτούμε. Η τρίτη τροπολογία μου αφορά το, την τροπολογία 8 στο άρθρο 12 όπου δίνεται στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να αφαιρέσουν τα φορολογικά ωφελήματα σε άτομα τα οποία είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη και πληρώνουν φόρους. Μα πώς είναι δυνατόν να έχουν όλες τις υποχρεώσεις του φορολογούμενου, αλλά να μην έχουν τα ωφέλη τα οποία δίνονται στους ηθαγενείς φορολογούμενους. Και αυτό μου φαίνεται ότι είναι σκληρό και απάνθρωπο και δεν έχει την παραμικρή δικαιολογία. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, και νομίζω ότι και αυτό θα μπορέσει να επιληθεί το τελευταίο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συζήτηση σε νομικό επίπεδο με την Κομισιόν. Η τροπολογία μου 4 λέει ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι αποσπασμένοι, εκεί η πρόταση οδηγία επιτρέπει για αυτού του εργαζόμενου να μην υπάρχει ισότητα μεταχείριση. Εγώ νομίζω ότι μία από τις ερμηνείε αυτές που έχουμε είναι ότι όταν δύο εργαζόμενοι έχουν αποσπαστεί σε άλλο κράτος μέλος, επιτρέπει η οδηγία να μην υπάρχει ισότητα μεταχείριση. Αυτή είναι μια ερμηνεία που μπορεί να δοθεί. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό είναι παράλογο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχει μια τέτοια ερμηνεία. Μου λέει η Κομισιόν ότι αυτό δεν είναι ο στόχος της Κομισιόν. Απλώς η, με, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι έχουν τη δική τους οδηγία που ρυθμίζει τα νομικά θέματα. Αν έτσι εντάξει, εάν είναι σεβαστή η ισότητα εργασίας μέσω της οδηγίας αυτής, έχει καλώς. Αλλιώς όμως δεν συμφωνώ. Κλείνω κύριε Πρόεδρε. Έχουμε την ευκαιρία να αρχίσουμε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Συμβουλίο και να εγκρίνουμε αυτό το έγγραφο σε πρώτη ανάγνωση. Έχουμε λοιπόν ένα παράθυρο ευκαιρίας όπου μπορούμε όχι 100% ίσως, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της νομοθετικής διαδικασίας να το φέρουμε σε πέρας. Εγώ πέρα του ότι είμαι Ισπανός είμαι και Ευρωπαίος. Θα πρέπει λοιπόν για μένα να είναι σαφές ότι θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια να κλείσουμε αυτό το θέμα σε πρώτη ανάγνωση αν το Συμβούλιο είναι έτοιμο να κινηθεί από τις θέσεις του. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ κατά 100% την θέση που είναι <clears throat> η θέση της πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Πρέπει να μάθει το Συμβούλιο και η Κομισιόν ακόμα ότι υπάρχουν δύο νομοθετικά σώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ακούσουν και τα επιχειρήματα του Κοινοβουλίου. Αν έχουν δίκιο, εγώ είμαι έτοιμο να αποδεχθώ αυτό το οποίο λένε. Αλλά αν έχει δίκιο το Κοινοβούλιο, θα πρέπει και το Συμβούλιο και η Κομισιόν να έχουν ανοιχτό πνεύμα για μια λύση συμβιβαστική ώστε να βρούμε κοινά στοιχεία, ιδίω για αυτά τα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπου διακυβεύεται και η ίδια η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακυβεύονται όλα αυτά που έχουμε πει τόσες πολλές φορές ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι χώρος παράνομης μετανάστευσης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα έρχονται εδώ πέρα με χαρτιά, με νόμιμο τρόπο αλλά συγχρόνω θέλουμε αυτά τα άτομα να ενσωματωθούν στην κοινωνία μα. Πρέπει να του δώσουμε όμω τα εργαλεία για να μπορέσουν να ενσωματωθούν. Δεν μπορούμε να έχουμε πολίτε πρώτη και δεύτερη κατηγορία λόγω τη φυλή του, του χρώματο του ή οτιδήποτε τέτοιο. Αν ενόμιμοι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα των ηθαγενών εργαζομένων, εκτό αν υπάρχει πραγματικά αποχρόν λόγο. Που αυτή τη στιγμή εγώ δεν τον διακρίνω σε το κείμενο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, κύριε Σιγητά. Ήσασταν πολύ δυναμικός και ορμητικός. Βασικά δεν έχουμε χρόνο. Αλλά οι μας δίνουν 10 λεφτά. Έχω τρεις ομιλητές που να πάρουν το λόγο. Ας τους ακούσουμε. Τι θέλετε, να κλείσουμε τη συζήτηση εδώ και να συνεχίσουμε αύριο ή να περιορίσω το χρονομιλία σας. Ό,τι θέλετε. Αύριο. Εντάξει, δέκα λεφτά θα ακούσουμε τώρα και θα τελειώσουμε αύριο. Κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Ο συνάδελφος κύριος Θέρκας ε, ξέρει πολύ καλά ότι συχνά συντάσσομαι μαζί του. Και εδώ συμφωνώ με το σημείο αφετηρίας του σε γενικές γραμμές. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ προσπαθούμε να εισαγάγουμε ένα νέο δικαίωμα. Ένα νέο είδος δικαιώματος. Και μία από τις πολιτικές που δεν θίγει, αν εξετάσουμε, αν λάβουμε υπόψη με το Συμβούλιο το, συγγνώμη, το, τον κανονισμό του 2003 του Συμβουλίου αναφέρεται σε ένα παράρτημα στις ειδικέ διατάξεις. Και αυτό το σημείο ο συνάδελφος δεν το φύγει. Εγώ θέλω να φύγει αυτό το παράρτημα για τις ειδικέ συνθήκες. Αυτό το σημείο δεν συμφωνούμε με τον Θέρκας. Και αυτό είναι νομίζω πολιτικό ζήτημα. Τώρα θα περάσω στις τροπολογίες για το εκτιμώντας 9, για την αιτιολογική σκέψη 9. Έχω την εντύπωση ότι το κείμενο της Κομισιόν είναι καλύτερο από του συναδέλφου μας, του κυρίου, του κυρίου Θέρκας. Η τροπολογία 2. Λέει ότι εντάσσονται στην οδηγία και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Κύριε Θέρκας, τι θέλετε να πετύχετε με αυτή τη νέα έννοια για, τους για τη διασυνοριακή μετακίνηση των εργαζομένων. Επίσης, Λέτε ότι δεν θα πρέπει να δοθούν άλλα δικαιώματα, αλλά να εφαρμοστούν αυτά τα δικαιώματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην τροπολογία 4, θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι συνέπειες από την κατάργηση του σημείου που προτείνεται για τις τροπολογίες 5 και 6, υπάρχει πρόβλημα με τη διατύπωση. Εκπαίδευση, κατάρτιση. Αυτά τα δύο θέματα νομίζω ότι εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογή της πρότασης. Μετά μιλάτε για τους, την εθνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την κοινωνική πρόνοια και κοινωνική προστασία. Αν με αυτή τη διαδικασία καταλήγουμε ε, σε μια πρόταση οδηγίας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια όρια. Στην τροπολογία 10... Μα ζητάτε να μην περιορίσουμε τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων αυτών. Δεν καταλαβαίνω ποιες είναι οι συνέπειες τροπολογίας 11. Γιατί 14 και 15 συμφωνώ. Υπάρχουν ε, στοιχεία τα οποία εγώ δεν δέχομαι και υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν στην ε, έκθεση, αλλά δεν, τα έχετε. Αυτά είναι τα σημεία διαφωνίας. Ο Τζιν Λάμπερτ ξέρει ότι υπάρχει μια τροπολογία περσινή η οποία είχε απορριφθεί επί τις οποίες εμείς συμφωνούσαμε. Αυτά ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστώ. Κύριε Σαγιά και Λάμπερτ στη συνέχεια. Tämän direktiivin päätarkoitus, aivan niin kuin esittelijä sanoi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, η οδηγία αυτή για αυτή την άδεια εγκατάσταση διαμονή εργασίας. Είναι σημαντικό να το δούμε στη συνέχεια εδώ. Ο εισηγητή πιστεύει ότι δεν υπάρχει πια αυτό το στοιχείο της αλληλεγγύη. Δεν νομίζω ότι είναι κατά της αρχή αλληλεγγύης. Νομίζω ότι εδώ δημιουργείται ένα μέσο για να δώσουμε τη μάχη μας πάνω σε αυτό. Αυτό το άρθρο το 12 νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα και υπάρχει ακόμα ευρύτερο δικαίωμα κοινωνικό χάρη σε αυτή την νέα διαδικασία και γι' αυτό θα έχει να κάνει με άτομα που διαθέτουν άδεια εργασίας και ταυτόχρονα άδεια διαμονής. Αυτό το σημείο είναι σημαντικό. Η Φινλανδία. Όλα αυτά βασίζονται στην άδεια διαμονής και η οδηγία εκεί που βασίζεται τι σημαίνει, τι συνεπάγεται ότι οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες είναι και σε άτομα που δεν έχουν ε, άδεια διαμονής αλλά για σύντομο χρονικό διάστημα διαμένουν εκεί και ένα, ένα κράτο μέλος. Τι γίνεται, πώς το αναγνωρίζει αυτό, όπως στη Φιλανδία πάνω χάρη έχουμε χίλια χιλιόμετρα σύνορα με τη Ρωσία και προέρχονται αυτοί οι εργαζόμενοι από τρίτη χώρα. Αν είναι μια Ρωσίδα εργαζόμενη θα έπρεπε να ζητήσει άδεια εργασίας σύντομης χρονικός διάρκειας για να έχει τη σχετική βίζα για να μπει και οι δικοί της στην οικογένειά της θα συνεχίσουν να ζουν στη Ρωσία αλλά χάρη σε αυτή την ε, αδειά ε, θα μπορούσαμε να έχουν, θα μπορούσαν να έχουν όλες αυτές τις υπηρεσίες από την Φιλανδία, ανεξάρτητα από το μισθό τους, από το εισόδημα τους. Τι θα γίνει όμως στο κάτω πώ ε, θα ζούσαν ε, εδώ εντάξει για όλα αυτά η Φινλανδία είναι κατά της οδηγίας αυτής. Και ακόμη κάτι, όπως το λέω, βασίζεται στην αρχή της διαμονής στη χώρα. Και δεν ξέρω αν έχει συλλογιστεί κανείς το κόστος όλων αυτών, γιατί μιλάμε, αναφερόμαστε σε 1.300.000 ευρώ κόστος. Εδώ στην τροπολογία 13 θα πρέπει σοβαρά να την εξετάσουμε γιατί αναφέρουμε σε άτομα που δεν εργάζονται. Τι έγινε τότε μας διαφεύγει η κατάσταση από τα χέρια. Θα υπάρχει μια διάσταση Αυτά και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. 7 παρά 20. Να διακόψουμε όμως εδώ, αυτό προτείνω, στο σημείο αυτό, έτσι, γιατί έχουμε ακόμα δύο μιλητέ και δεν θα ήταν δίκαιο να του παίρνουμε τόσο πολύ χρονομιλίες. Αύριο πρώτο σημείο να εξεταστεί αυτό στη μεσιά μα διάταξη και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Λάμπερτ που ελπίζουμε να είναι εδώ και κυρία η εδώ Ελπίζουμε να είναι παρούσοι και οι δύο και έτσι να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Αυτά και σας ευχαριστώ.